Καλησπέρα συνάδελφοι. Ε, ε, σας καλωσορίσω στην ε, κοινή αυτή, στο κοινό αυτό εργαστήριο ε, της Επιτροπής Προπολογισμών με την Επιτροπή ΕΚΟΝ για την δημοσιονομική ικανότητα, για την ενίσχυση και διεύρυνση της Ευρωζώνης. Είναι ένα θέμα όπου οι επιτροπές μας έχουν ε, κάνει πολλή δουλειά τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά υπό την αιγίδα και κατεύθυνση της Περδάνς ε, Μπερές ε, και τον κύριο Μπέγκε από τη δική μας επιτροπή. Η κυρία ε, Μπερές είναι από την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Και θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε και να σταθεροποιούμε το κοινό μας νόμισμα. Υπήρχε και μια πλειοψηφία υπέρ της έκθεσης Μπερές Μπέγκε στην Ολομέλεια πέρσι το Μάρτιο όταν υιοθετήθηκε αυτή η έκθεση. Επίση, έχουμε ένα μακρύ κατάλογο από πολύ διακεκριμένους ομιλητέ. Σήμερα το απόγευμα θα ξεκινήσουμε με τους δύο εισηγητές που θα κάνουν κάποιες αγωγικέ παρατηρήσεις και μετά ε, θα πάρουμε τους ομιλητές ένα προς ένα πριν δώσουμε στους εισηγητές στην, ε, που είναι η κυρία Μπερές και ο κύριος Μπέγκε, αλλά πρώτα θα δώσω το λόγο στον συμπρόεδρο, ε, πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, τον κύριο Γουαλτιέρη. Χαίρομαι που διοργανώσαμε αυτό το κοινό εργαστήρι των δύο επιτροπών για τη δημοσιονομική ικανότητα πρέπει την ενίσχυση και διεύρυνση της Ευρωζώνης, επιτροπές ΕΚΟΝ και BUDGE, που συνεργάστηκαν με πολύ παραγωγικό τρόπο, όπως όλοι ξέρουμε. Έχουμε και τους δύο συνεισηγητές, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν τη δουλειά που κάναμε, θα μας κάνουν μια αρχική εισαγωγή με βάση τα όσα λέει η δική μας έκθεση και με βάση την εργασία που παρουσίασε στο μεταξύ κομισιών και όσα θα παρουσιάσει εφ' εξής, θα μπούμε λιγάκι στην ουσία του θέματος. Μιλάμε για πτυχές της ΟΝΕ και δημοσιονομικές πτυχές. Έχουμε, ας πούμε, παντρέψει αυτές τις δύο πτυχές, ε, ψάχνουμε την τομή τους, θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε από κοινού, ούτω ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε μια κατάλληλη απάντηση στα προβλήματα και να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις στα προβλήματα της ΟΝΕ. Και στον προβληματισμό που γίνεται για τον προπολογισμό μας. Πρόκειται λοιπόν για μια πολύ επίκαιρη συζήτηση στα πλαίσια αυτού του εργαστηρίου. Ευχαριστώ εκ των προτέρων του ομιλητέ για την παρουσία του. Θα μπούμε σε διάφορα θέματα, πολύ σημαντικά, και ελπίζω ότι αυτά θα μας βοηθήσουν να δώσουμε μια συνολική απάντηση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε διάφορα επιμέρους νομοθετικά ζητήματα. Uh, Συνεπή τρόπο, ούτως ώστε να σημειωθεί συγκεκριμένη πρόοδος. Με σκοπό βέβαια την καλύτερη διακυβέρνηση. Δεν θέλουμε να ολοκληρώσουμε απλώς στην ΟΝΕ. Θέλουμε να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα για να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά μας και να εξασφαλίσουμε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο διακυβέρνησης της Ευρωζώνης. Η Περβάνς Μπερέση έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Περβάνς. Ευχαριστώ. Συμπρόεδρε. Δυόμιση λεφτά μου δίνετε για να παρουσιάσω αυτό το θέμα. Τι να πω, είναι πολύ λίγο. πάρα πολύ. Να σας υπενθυμίσω ποια ήταν η θέση που υιοθετήθηκε από το Κοινοβούλιο. Όταν εξετάσαμε την έκθεση Μπερές Μπέγκε. Ε, θα διαβάσω τρεις παραγράφους. Στην πρώτη παράγραφο λέμε ότι η δημοσιονομική ικανότητα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει το, ε, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και επιπλέον δυναμικό δημοσιονομικό δυναμικό για την Ευρωζώνη. Μιλάμε ξεκάθαρα για την μετεξέλιξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα στα πλαίσια του συνολικού προπολογισμού και τη Ευρωζώνη. Εν συνεχεία, λέμε ότι ο μηχανισμό σταθερότητα θα εκπληρώνει βεβαίω τα δικά του καθήκοντα, αλλά θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω και να γίνει ε, ε, ένα ενίο ένα νομισματικό ταμείο ούτω ώστε να έχει ικανότητα χρηματοδότησης για να απορροφά τα συμμετρικά και ασύμετρα σοκ. Είμαστε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο. Αυτή είναι η πιθανή εξέλιξη. Έχουμε τις σημερινές λειτουργίες και μιλάμε για την στήριξη που μπορεί να δώσει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για, πρα, για να αποκτήσουμε πράγματα που λείπουν από την ονέ μας και να τη σταθεροποιήσουμε. Τέλο, λέμε, η σταθεροποίηση γίνεται μέσα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό σταθερότητα και το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Θα πρέπει να συμπληρώνεται από κατάλληλου μηχανισμού απορρόφησης των σοκ. Αυτά είναι τα στοιχεία που είχαμε πει στην εκθεσή μα. Επ' αυτή τη βάση η πρόταση τη Κομισιόν σημειώνει ότι θέλουμε να μετασχηματίσουμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό σταθερότητα και να τον βάλουμε στο, ε, στο κοινοτικό πλαίσιο δυνάμει του άρθρου 352, αλλά ξέρετε ότι προς το παρόν το Κοινοβούλιο δεν εντάσσεται σε αυτόν τον κύκλο, γιατί το Συμβούλιο συζητάει σε τεχνικό επίπεδο για την αντίληψη που έχει για την ε, μελλοντική μορφή του μηχανισμού σταθερότητας και το Κοινοβούλιο θα πει απλώς ναι ή όχι. Έχει δυνατότητα δηλαδή έκδοσης σύμφωνης γνώμης. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι έχει πολύ νόημα αυτό το εργαστήρι, υπό τον όρο βεβαίω ότι θα κάνουμε και συγκεκριμένε προτάσει. Τώρα, επί τη ουσία. Euh, ε, ελπίζουμε ότι θα μετασχηματιστεί αυτό ο μηχανισμό σταθερότητα, το ελπίζουμε και το θέλουμε. Πέρα από αυτά που γράφει η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, και στις απόψεις των άλλων βεβαίως, θέλουμε να διασταυρώσουμε ότι η καλή φόρμουλα είναι η ενσωμάτωση, η ένταξη στο κοινωνικό, κοινωτικό πλαίσιο και αυτή η μετατροπή του μηχανισμού σταθερότητα να μην το αδειάσει από το νόημά του, να μην αφαιρέσει αρμοδιότητες από την Κομισιόν στο θέμα της δημοσιονομική εποπτείας, που είναι η αρμοδιότητα προς το παρόν της Κομισιόν, και ο Ευρωπαϊκό ε, Μηχανισμό Σταθερότητα θα μετασχηματιστεί σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, αλλά αυτό να μην γίνει πρόσχημα το οποίο θα οδηγεί σε διαβουλεύσεις ε, τύπου άρθρου 4 ε, και αφαιρέσει αρμοδιότητες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τρίτο σημείο που θέλω να υπενθυμίσω. Αυτός ο μετασχηματισμός του μηχανισμού σταθερότητας, αλλά εντάξει αυτό θα συζητηθεί σε πολιτικό επίπεδο, ε, σε μία αυτόματη αναδιάρθρωση του χρέου, να μην οδηγήσει σε αυτό. Γιατί αντί να λύσουμε ένα πρόβλημα, θα λύσουμε ένα μένα, θα δημιουργήσουμε ένα καινούριο. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να συνοδευτούν από μετασχηματισμού στο επίπεδο τη διακυβέρνηση. Δεν έχω χρόνο να μπω σε αυτό όμω. Απλώ ένα ερώτημα θέλω να θέσω. Πώ βλέπετε την εξέλιξη τη διακυβέρνηση αυτού του μηχανισμού σταθερότητα και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο επίπεδο αυτό. Και τελευταίο σημείο που θα με υπενθυμίσω είναι ότι μεταξύ των νέων αρμοδιοτήτων αυτό το νέο ταμείο ας πούμε θα μπορούσε να είναι και ένα δίχτυ ασφαλείας στο δεύτερο πυλώνα της α, ε, Τραπεζικής Ένωσης. Δηλαδή ένα νέος, ένας νέος μηχανισμός στήριξης για τον τρίτο πυλώνα, δηλαδή για την εγγύηση των καταθέσεων. Αυτό λοιπόν θα είναι σημαντικό για, ε, σημείο για μας και πρέπει να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Μπέγκε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω όσα είπε η συνάδελφός μου η Υπερβάνς Μπερές ως εισαγωγή. Απλά θα συμπληρώσω με παρατηρήσεις. Πολύ απλά. Ένα χρόνο πριν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίθηκε η έκθεση για τη δημοσιονομική ε, δυνατότητα. Υπήρξε πολλή δουλειά που είχε προηγηθεί βέβαια, πολλές ακροάσεις. Δεν υπήρξε <coughs> πρόβλημα στις, ε, στην ψηφοφορία. Είχαμε ακούσει ήδη τις προτάσεις Μακρό για την ε, προβλεπτική οικονομική διαχείριση ε, και σίγουρα οι πολίτες μας έχουν ε, την αξίωση να συζητηθούν προτάσεις και να εγκριθούν προτάσεις που θα οδηγούν γενικά σε μεγαλύτερη ασφάλεια οικονομική και κοινωνική σε ένα κόσμο που φαίνεται να είναι ασταθής και ρευστός. Δηλαδή η σταθεροποίηση της οικονομίας και η σταθεροποίηση της ΩΝΕ είναι το βασικό ε, ζήτημα. Έχουμε το πακέτο της Κομισιόν και υπήρξαν ε, στην ε, νέα συνθήκη του νέου μεγάλου σας στη Γερμανία κάποιες ε, ενδιαφέρουσες διατυπώσεις κάτι που δεν είχαμε ακούσει παραδείγματο χάρη εδώ και ένα χρόνο, ενίσχυση των οικονομικών της Ένωση, δημοσιονομική ενίσχυση, σύγκληση ε, και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρωζώνη πρέπει να υποστηριχθούν ή επίσης ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός ε, Σταθερότητας πρέπει να μετατραπεί σε ένα ελεγχόμενο από το Κοινοβούλιο ε, νομισματικό ταμείο και επίσης τα δικαιώματα των εθνικών κοινοβουλίων παραμένουν αναπαλωτρίωτα. Οι Υπουργοί Οικονομικών ε, δείχνουν να είναι επιφυλακτικοί. Δεν έχει βέβαια απόλυτα σχέση με το σημερινό θέμα, αλλά πρέπει να βρούμε απαντήσεις. Ε, ο Γιάνν Ολμπρίχτ, που είναι συγητής μας για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, υπάρχουν ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα και την ασφάλεια. Και έχουν να κάνουν αυτά τα θέματα σίγουρα και με τη δημοσιονομική ικανότητα. Πώς ε, θα αποφύγουμε δηλαδή ένα λάθος Έχουμε τη συνοχή, αλλά δεν θα πρέπει να την αντιπαραβάλλουμε με την πολιτική ασφάλειας ε, ή την εξωτερική πολιτική ή έχουμε την προστασία συνόρων από τη μία και την πολιτική γειτονία από την άλλη. Δεν πρέπει το ένα να είναι αντίθετο ε, προ το άλλο. Θέλουμε ένα πακέτο, τέσσερα-πέντε σημεία, στα οποία πρέπει να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη, πάντα στο πλαίσιο αυτή τη ασφάλεια, αλλά ένα μέρο του πακέτου θα πρέπει να είναι βιώσιμη σταθεροποίηση του ευρώ, τη οικονομία και της Νομισματικής Ένωσης. Αλλά χωρίς να θέλουμε να περιθωριοποιήσουμε κάποιο κράτος μέλος. Αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη. Και σε ό,τι αφορά το government structure, είναι ένα θέμα το οποίο το συζητήσαμε και ένα θέλω να πω, επειδή ε, υπάρχει αυτή η διατύπωση που μιλάει για κοινοβουλευτικό έλεγχο όταν δημιουργήθηκε το EFSM ήταν 60 δις, ε, αυτά τα οποία εκεί κρατών και κυβερνήσεων μέσα στους ιδίους πόρους. Αλλά αυτό έγινε χωρίς ε, καμία ε, γνωμοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί γιατί έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαιώματα, έχει αρμοδιότητε. Θα περιμένω και εγώ να ακούσω τι θα πούνε εμπειρογνώμε. Θέλουμε να έχουμε μια δομή εφτάκτη και ίσω ε, πιο σταθερή σε εσύ. Με το άρθρο 122 που είχαμε χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα. Ελπίζω το σημερινό εργαστήριο να δώσει ε, κάποιες σκέψεις ε, στα ερωτήματα αυτά που θα απασχολήσουν το πολιτικό μας έργο στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο συνεισηγητές. Σημαντικές οι παρατηρήσεις και η τελευταία Δηλαδή ε, δεν ε, θα είναι παρακρίμα να έχουμε ένα εντελώς άτολμο νέο εργαλείο, το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή που δεν θα έχει επαρκή προπολογισμό. Ελπίζω οι δικοί μας να μας βοηθήσουν να δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα και προβλήματα αυτά που έθεσαν οι δύο εισηγητέ. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τον κύριο Κλάου Ρέγκλινγκ, τον διευθύντη του ESM, Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ που με καλέσατε. Χαίρομαι πάντα να βρίσκομαι στο Ευρωκοινοβούλιο για ανταλλήγη απόψεων. Το σημερινό θέμα είναι σημαντικό. Οι δημοσιονομικές πτυχές της εμπάθυνσης της της Ένωση. είναι σημαντικό, είναι και επίμαχο το θέμα αυτό στα κράτη-μέλη μας. Και πρώτο ξεκινήσω στην ουσία του θέματος. Θα ήθελα να πω ότι είμαι τακτικό επισκέπτη εδώ παρόλο που δεν υπάρχουν επίσημοι δεσμοί ανάμεσα στο ESM και στο Ευρωκοινοβούλιο, ο δικός μου θεσμός λογοδοτεί στις χώρες της Ευρωζώνης, ε, των οποίων οι χρηματικές συνεισφορές μας επιτρέπουν να κάνουν τη δουλειά μας. Από δική μου άποψη δεν υπάρχει έλλειμμα λογοδοσίας ή δημοκρατίας, αλλά είναι μια άποψη που δεν την μοιράζονται όλοι. Οι 19, τα 19 μέλη του ΔΣ, οι Υπουργοί Οικονομικών, που είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ESM, λογοδοτούν στα δικά του εθνικά κοινοβούλια. Αλλά είναι πολύ καλή πρακτική αυτή η ανταλλαγή απόψεων εδώ, σε αυτό το σώμα, ιδιαίτερα τώρα που δουλεύουμε προς τον κοινό στόχο του να φτιάξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, την νομισματική ένωση πιο ισχυρή και την οικονομία πιο ανθεκτική. Το πακέτο του Δεκέμβρη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέβλεπε, ε, μάλλον έδωσε ένα, μια όθηση στην εμπάθηση της Νομισματικής Ένωσης. Στόχος είναι να ε, αποκαταστήσει κάποιες σημαντικές αδυναμίες στη σύσταση της Νομισματικής Ένωσης, κάτι το οποίο καλωσορίζω θερμά. Έχει ξεκινήσει τώρα το έργο στα δύο θέματα όπου υπάρχει συνένεση, ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και ε, μεταξέλιξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, ε, ε, του ESM. Τα δημοσιονομικά μέσα είναι ένα άλλο σκέλος της συζήτησης, αλλά δεν μπορούμε να τα βλέπουμε σε απομόνωση. Η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και η αξιοποίηση νέων δημοσιονομικών εργαλείων εξυπηρετούν ακριβώς τον ίδιο οικονομικό στόχο, δηλαδή την αύξηση του επιμερισμού, του οικονομικού κινδύνου μέσα στην Νομισματική Ένωση. Υπάρχει όμως και ένα αντάλλαγμα ανάμεσα στα δύο. Όσο πιο μεγάλος κίνδυνος επιμερίζεται ε, ανάμεσα στο ιδιωτικό τομέα, τόσο λιγότερη ανάγκη υπάρχει να γίνει επιμερισμός των κινδύνων από τα δημοσιονομικά εργαλεία θα ε, πρέπει να δούμε το πακέτο στην ολοτητά του, ε, γιατί ε, υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις για τα δημοσιονομικά μέτρα και θα πάρει χρόνο μέχρι να επιτευχθεί κάποια συμφωνία. Προτού δούμε τώρα τις δημοσιονομικές πτυχίες, θα ήθελα να δω τους δύο τομείς του έργου της εμβάθυνσης της Νομισματικής Ένωσης, όπου υπάρχει κάποια σύγκληση. Σε ό,τι φορά την Τραπεζική Ένωση, η Ευρώπη έχει ήδη θεσπίσει τους δύο πρώτους πυλώνες, ε, τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, το SSM και το ενιαίο ταμείο εξυγένσης, το SRF. Για να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση, το SRF χρειάζεται ένα backstop, ένα δίκτυο χρηματοπιστωτικής προστασίας ένα κοινό σύστημα εγγύηση των καταθέσεων είναι ένα σημαντικό βήμα, διότι θα προωθήσει την χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση και την εμπιστοσύνη ανάμεσα στου καταθέτε. Γνωρίζουμε όμω ότι αυτό είναι πολιτικό επίμαχο θέμα, διότι υπάρχουν κάποια υφιστάμενα παλαιότερα προβλήματα σε τράπεζε ή σε κάποια τραπεζικά συστήματα, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αλλά ε, δεν αμφισβητείται ο απότερο στόχο μα. Στο θέμα τη μεταξέλιξη του δικού μου θεσμού θα ήθελα να πω ότι όταν ακούω τι συζητήσει στο Eurogroup ε, νιώθω ότι υπάρχει ε, στήριξη ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης για τη μεταξέλιξη του ESM ε σε ένα πλήρως οργανωμένο μηχανισμό σταθεροποίηση στήριξης. Ένα, ε, ένας πιο ισχυρό ESM δεν είναι ένας στόχο από μόνο του, αλλά όπως και με την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωση, μπορεί να είναι ένα στοιχείο που θα κάνει την νομισματική ένωση λιγότερο τρωτή και θα δείξει ότι η Ευρώπη αναλαμβάνει περισσότερη ευθύνη για να επιλύσει τα δικά της προβλήματα. Εκτός από το δίκτυο προστασίας για το SRF, το ESM θα παίξει ένα ευρύτερο ρόλο σε, οποιαδήποτε μελλοντικά προγράμματα ε, χρηματοοικονομικής βοήθειας. Μαζί με την Επιτροπή θα είναι από κοινού αρμόδιο για το σχεδιασμό, τη διαπραγμάτευση και την παρακολούθηση νέων προγραμμάτων. Βέβαια, αυτή η συνεργασία θα πρέπει βέβαια να ε, τηρεί τις αρμοδιότητες της Επιτροπής και δεν πρέπει να υπάρχει επικάλυψη έργου. Το ESM θα μπορούσε να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις για μελλοντικές αναδιαρθρώσεις του δημοσίου χρέους, έτσι ώστε να γίνουν πιο συστηματικές αυτές οι διαπραγματεύσεις και πιο προβλέψιμες παρά στο παρελθόν. Θα έχει και μια, ένα νέο δημοσιονικό μέσο μακροοικονομικής σταθεροποίησης ή προστασίας των επενδύσεων. Και έρχομαι τώρα στο κύριο θέμα της ημέρας, τις δημοσιονομικές πτυχές της εμβάθυνσης της Νομισματικής Ένωσης. Για να καταλάβουμε καλύτερα πώς το βλέπω εγώ το θέμα, θα ήθελα να συζητήσω πρώτα απ' όλα αυτό τον επιμερισμό του οικονομικού κινδύνου. Ο, αυτός ο επιμερισμός του οικονομικού κινδύνου δεν είναι αναπτυγμένο στην Ευρωζώνη όταν το συγκρίνουμε με τις ΗΠΑ, αλλά και με τον επιμερισμό του κινδύνου στη Γαλλία ή και στη Γερμανία σε εθνικό επίπεδο. Στις ΗΠΑ, αν ε, υπάρχει ένα σοκ που πλήττει μια πολιτεία ή μια ομάδα πολιτιών, αυτό μεταδίδεται πιο εύκολα σε όλη τη χώρα παρά στην Ευρωζώνη. Σημαίνει ότι αυτά τα σοκ μπορεί να είναι πιο επώδυνα στην Ευρώπη. Ε, ιδιαίτερα γιατί η νομισματική πολιτική στην ναι, δεν είναι και διαθέσιμη για να αντιμετωπίσει προβλήματα της κάθε χώρας. Η αύξηση του, του επιμερισμού του κινδύνου θα μπορούσε να προλάβει ε, το, το λίστημα μιας χώρας σε πιο σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Δηλαδή αυτό θα μας κάνει λιγότερο ευάλωτους. Στη ΣΥΠΑ, αλλά και εντός της Γαλλίας ή της Γερμανίας, ο επιμερισμός του κινδύνου σε μεγάλο βαθμό γίνεται μέσα στον ιδιωτικό τομέα, μέσα από τις τράπεζες, τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τις ροές των κεφαλαίων. Αλλά οι χρηματοπιστωτικές αγορές της Ευρώπης είναι ακόμη κατακαιρματισμένες ε, γι' αυτό και η ε, ε, ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης θα πρέπει να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα στην εμπάθεση της Νομισματικής Ένωσης. Η, επίσης, ε, η συνέχιση του έργου της Ένωσης των Κεφαλογορών θα είναι σημαντική επιπρόσθετη βελτίωση. Τα δημοσιονομικά εργαλεία βοηθούν στην πρόθεση του επιμερισμού του κινδύνου, παρόλο που ε, δεν χρειάζονται τόσο, τόσο, τόσο πολύ ε, εάν ο επιμερισμός του κινδύνου μέσα από τις αγορές λειτουργεί καλά. Υπάρχουν πολλά ε, στοιχεία στον δημοσιονομικό χώρο τα οποία μπορεί να μην χρειαζόμαστε για μια σωστή λειτουργία της νομισματικής ένωσης. Δεν χρειαζόμαστε ούτε μεγαλύτερα επιπρόσθετα, ε, μεγαλύτερες επιπρόσθετες μεταφορές κονδυλίων ανάμεσα σε χώρες. Ε, ακόμη και εάν είναι μικρός ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, μόνο 1% του ΑΕΠ ε, οι φτωχότερες χώρες ε, ήδη λαμβάνουν κονδύλια από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που μπορεί να είναι στο 4% του μεγέθους της οικονομίας τους που είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Εκτός αυτού, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το σχέδιο Juncker ήδη περιέχουν κονδύλια για την πρόθεση επενδύσεων. Ε, Επίσης δεν χρειαζόμαστε επιπρόσθετα μέτρα και μέσα αντιμετώπισης των μεγάλων συμμετρικών σοκ που πλήττουν την περιφέρεια. Οι δημοσιονομικοί κανόνες ήδη επιτρέπουν συγχρονισμένη δαπάνη του προπολογισμού. Ε, αυτό το περιθώριο χειρισμού αξιοποιήθηκε με επιτυχία ε, σε ανταπόκριση στις κρίσεις του 2009 και του 2010 και ε, εκεί η ΕΚΤ επίση ε, θα βοηθήσει αν υπάρχει μεγάλο συμμετρικό σοκ. Εκεί που βλέπω ότι υπάρχει ένα σημαντικό χάσμα στα δημοσιονομικά εργαλεία είναι όταν μία κρίση δεν πλήττει όλη την περιφέρεια, αλλά μόνο μία ή δύο χώρε. Τα λεγόμενα σύμμετρα σοκ. Έχω δώσει και ελπίζω το υποθετικό παράδειγμα της Ιρλανδίας, εάν ε, θα την έπλητε ε, ε, το Brexit σε μεγάλο βαθμό. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να στηρίξει τη χώρα. Όταν σκεφτούμε τις δημοσιονομικές πτυχές της εμβάθυνσης της Νομισματικής Ένωσης, μια νέα δημοσιονομική δυνατότητα μακροοικονομικής σταθεροποίησης θα πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα. Θα πρέπει να είναι σημαντικός διάβλος για δικτύων επιμερισμό των κινδύνων. Αυτό το εργαλείο μπορεί να σχεδιαστεί χωρίς αμοιβαία κάλυψη του χρέους και χωρίς να δημιουργηθούν μόνιμες μεταφορές κονδυλίων. Παραδείγματα στη ΣΥΠΑ, όπως τα Rainy Day Funds, τα ταμεία για τις άσχημες μέρες ή ένα συμπληρωματικό σχέδιο ανεργίας. Η το, το μέσο αυτό θα πρέπει να έχει τη μορφή ενός ανανεώσιμου ταμείου, όχι ενός ετήσιου προϋπολογισμού και θα πρέπει να αποπληρώνεται εντός ενός οικονομικού κύκλου, δηλαδή 5-6 χρόνια. Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια του EMS θα μπορούσαν να ήταν μια δυνατότητα για ένα τέτοιο μέσο που να συνδέεται με μια ελαφρύτερη με ελαφρύτερες προϋποθέσεις αυτά τα ε, δάνεια θα μπορούσαν να διατίθενται για σταθεροποίηση των επενδύσεων, αν υπάρχει ε, κάποια κρίση. Υπάρχουν και άλλες ιδέες σχετικά με τις δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνουν τον προπολογισμό ε, χρηματοδότηση από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη χρηματοδότηση των δημοσίων αγαθών όπως την προστασία εξωτερικών συνόρων θα ήταν χρήσιμο για σκοπούς αποδοτικότητας και πίζω να το εξετάσετε στα πλαίσια του επόμενου πιδελταπή. Η αναμόρφωση των δημοσιονομικών κανόνων επίσης μελετώνται. Ήταν στην αρχή εύκολη, ευκατανόητη, αλλά από τότε, από την αρχή της ΟΝΕ έχουν τώρα γίνει πολύ περίπλοκοι και δύσκολοι ακόμη και για τους εμπειρογνώμονες. Τέλος, θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει ένας Υπουργός ε, Οικονομικών Ευρωζώνης ε, εάν υπάρχει ένας προπολογισμό της Ευρωζώνης και για σκοπούς συντονισμού και για σκοπούς εκπροσώπησης. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι είμαι σίγουρο ότι η Ευρώπη μπορεί να αναλάβει κάποια σημαντικά ε, μέτρα φέτος για να κάνει την νομισματική ένωση πιο ισχυρή και να, να προστατεύσει περισσότερο τους πολίτες κατά το αντίκτυπο ενός επικειμενού σοκ. Για μένα ως οικονομολόγο το όφελος θα ήταν ότι η Ευρωζώνη θα απολαμβάνει αυτό τον επιμερισμό των οικονομικών κινδύνων και αυτό μπορεί να γίνει κυρίως μέσω των αγορών αλλά και μέσω της επιλογής επιπρόσθετων μέσων και εργαλείων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για παρατηρήσεις. Τι σημαίνει αυτό το predictable, το προβλέψιμο που είπατε. Θα σας ρωτήσω αργότερα όμως. Πάμε τώρα στην κυρία Νιές Μπενασί Κερέ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με προσκαλέσατε γιατί συμμετείχα σε αυτό το γαλλογερμανικό γκρουπ με 14 εμπειρογνώμονε που έπρεπε να κάνει προτάσει για την Ευρωζώνη. Αυτό που θα κάνω στο λίγο χρόνο που μου δίνεται είναι να παρουσιάσω τρεις άξονες προτάσεων που θα πρέπει να αναλυθούν χωριστά πριν συνδυαστούν για να φτιάξουν ένα πακέτο. Το πρώτο είναι τα δημόσια αγαθά, ε, η σταθεροποίηση και η δημοσιονομική ευθύνη το τρίτο. Ας ξεκινήσουμε. Με τα δημόσια αγαθά. Ποιο είναι το πρόβλημα. Πάντα θα θέτω αυτό το ερώτημα και μετά ε, θα αναζητήσω τα εργαλεία για να επιληθεί το πρόβλημα. Λοιπόν, παραδοσιακά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα δημόσια αγαθά παράγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τον ενωσιακό προπολογισμό μεγάλο θέμα σήμερα. Τι θα πρέπει, θα πρέπει μάλλον να εμπλέξουμε την Ευρωζώνη ή το ενωσιακό επίπεδο, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως οι χώρες της ε, Ευρωζώνης έχουν διαφορές, διαφορετικές προτιμήσεις από τις χώρες που δεν συμμετέχουν στην Ευρωζώνη. Δεύτερον, η πολιτική οικονομία προφανώς είναι πολύ πιο εύκολο να συμφωνήσουν οι 19 από τους 27 ή θα μιλήσω για τη σταθεροποίηση, αλλά κάποιες χώρες είναι πιο ασταθείς από κάποιες, όλες, από κάποιες άλλες. Το να έχουμε τις ε, σταθερές χώρες ε, που θα χρηματοδοτήσουν ένα σύστημα ε, σταθεροποίηση για να το κάνουμε πρέπει να δώσουμε κάτι σε αντάλλαγμα. Και τέλος, είναι δυνατόν τα δημόσια αγαθά της Ευρωζώνης που εξασφαλίζουν την δημοσιονομική σταθερότητα, που είναι καλό για αυτές τις χώρες, Γι' αυτό υπάρχει μια δικαιολόγηση για την στήριξη του ενιαίου ταμείου εξυγίανσης και η σύγκληση μπορεί να θεωρηθεί δημόσιο αγαθό. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν ότι αποκλήσεις στις χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να οδηγήσουν σε έκρηξη. Λοιπόν, έχουμε την πρόταση της Κομισιόν μέσα από το πλαίσιο. Ε, μιλάει για την δημοσιονομική στήριξη του Ενιαίου Ταμείου Ξυγίνησης, μια υποστήριξη των χωρών ε, που θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωζώνη, υποστήριξη των ε, διαφορετικών μεταρρυθμίσεων για την οικονομική σύγκληση και ασφαλή στοιχεία ενεργητικού. Είναι ένα στοιχείο που εξασφαλεί σταθερότητα, οικονομική φυσικά σταθερότητα. Ποια είναι η πρότασή μας. Ε, 7 επί 7 λέγεται. Είναι επίσης δημοσιονομική στήριξη του SRF και του μελλοντικού EDIS, ε, του συστήματο εγγύηση των καταθέσεων και ασφαλή περιουσιακά στοιχεία ή στοιχεία ενεργητικού. Δεν μιλήσαμε για τη χρηματοδότηση άλλων δημοσίων αγαθών, όχι γιατί είμαστε αντίθετοι, αλλά γιατί θέλαμε να επικεντρωθούμε στου δύο, άλλου άξονε, που είναι η δημοσιονομική σταθεροποίηση και η δημοσιονομική ευθύνη. Δημοσιονομική σταθεροποίηση. Ποιο είναι το πρόβλημα. Έχουμε ασύμετρα σοκ και έχουμε και συμμετρικά σοκ. Καταρχά τα σύμμετρα. Υπάρχει μια, ένα χάσμα ανάμεσα σε δύο επίπεδα σταθεροποίηση. Έχουμε εθνική ε, δημοσιονομική σταθεροποίηση μέσα στο, στα πλαίσια του Συμφώνου ε, Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Για χώρε που έχουν μεγάλη κρίση, του δίνουμε δάνεια ε, τύπου ESM. Ε, από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα. Βεβαίω, κάποιε χώρε έχουν προθυμία για να ζητήσουν βοήθεια. Υπάρχει μια ανακολουθία ανάμεσα στα δύο, γιατί σε ορισμένε περιπτώσει μπορεί να υπάρχουν πολλά προβλήματα. Μερικές φορές έχουμε προβλήματα ρευστότητας και οι διάφορες χώρες δεν θέλουν να μπουν σε πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και πολλές ενδιάμεσες περιπτώσεις. Έχουμε τώρα τα συμμετρικά σοκ που είναι και τα περισσότερα στην Ευρωζώνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον. Ε, προς το παρόν δεν έχουμε συνολική δημοσιονομική αντιμετώπιση. Δεν υπάρχει δημοσιονομικό συντονισμός ε, και οι απόπειρε που έχουν γίνει έχουν αποτύχει, δεν υπάρχει κεντρικό προπολογισμό επίση. Αυτό που παρατηρήσαμε είναι το 2011, 2012 και 2013 είναι προκυκλικές πολιτικές και δεν υπάρχει κανένα τρόπο να αναγκάσει μια χώρα να κάνει πολιτικές αντικυκλικές και να συμμετάσχει σε συνολική προσπάθεια σταθεροποίησης. Αυτό το πρόβλημα ε, μπορεί να γίνει πιο οξύ στο μέλλον δεδομένη τη αύξηση ε, του επίπεδου του χρέου. Όταν έχει πολύ ψηλό επίπεδο και ε, ο λόγο χρέου προ ΑΕΠ, υπάρχει, μια χώρα, υπάρχει φόβος μια χώρα να διωχθεί από τις αγορές. Σε αυτό το πλαίσιο, ποια είναι η πρόταση της Κομισιόν, λοιπόν. Ε, δημοσιονομικό ε, δυναμικό. Δυνατότητα δανεισμού, αυτόματη ενεργοποίηση, ένα μείγμα δανείων και μεταφορών κονδυλίων, ε, σταθεροποίηση των επενδύσεων σε συμφωνία με τον ενωσιακό προπολογισμό. Επίση, προληπτική πιστοτική γραμμή από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα, μελλοντικό Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, πιθανώ ένα μηχανισμό ασφάλεια και αναθεώρηση των κανόνων των δημοσιονομικών. Ε, εμείς τι προτείνουμε, 7 επί 7. Ε, προληπτική δημοσιονομική γραμμή του ESM, ε, δημοσιονομική ικανότητα, ε, ένα ταμείο για τις ε, δύσκολες μέρες, ε, το, το 0,1% του ΑΕΠ, αυτόματη ενεργοποίηση, η προϋποθέση, η αιρεσιμότητα θα αφορούν τη χρήση του, των χρημάτων, το πώς θα, θα πρέπει τα χρήματα αυτά δηλαδή να δαπανηθούν, όχι να τα, να τα αποταμιεύσουν. Και δεν θα υπάρχει δυνατότητα δανεισμού. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σήμερα για να έχουμε κοινό δανεισμό και πιστεύουμε ότι σε περίπτωση που υπάρχει μια τεράστια κρίση που αφορά όλες τις χώρες της ε, Ευρω... Ευρωζώνης έχουμε ένα μηχανισμό στήριξης. Η μεταρρύθμιση του SGP με ένα κανόνα δανεισμού που αντικαθιστά το περίπλοκο πλαίσιο που έχουμε σήμερα. Ε, κανόνες δανεισμού πολύ πιο εύκολους, ε, πιο εύκολο να τα καταλάβουν οι εθνικοί βουλευτές και πιο εύκολο να τα παρακολουθήσουμε σε επίπεδο ευρωζώνης και πιο ε, ανοιχτό σε αντικυκλικές πολιτικές. Τέλος, δημοσιονομική ευθύνη. Ποιο είναι το πρόβλημα. Σήμερα έχουμε το εξής πρόβλημα. Θα θέλαμε να έχουμε ένα κανόνα ε, μη ε, διάσωσης και αυτός να είναι αξιόπιστος. Αλλά αν γίνει ε, αξιόπιστος μπορεί να δημιουργήσει το σύνδρομο Ντοβίλ, δηλαδή κίνδυνο κρίσης ομολόγων. Το status quo είναι ότι δεχόμαστε ότι η ρήτρα αυτή για μη διάσωση παραμένει μη αξιόπιστη. Σε περίπτωση που δεν έχουμε τελικό δανειστή σε επίπεδο ευρωζώνης, Είχαμε δηλαδή την ΕΚΤ και τα λοιπά, αλλά πάντα με πρόγραμμα. Δεν υπήρχε πραγματικό ε, τελικός δανειστής, για... υπήρχε για τις τράπεζες, αλλά όχι για τα κράτη. Σε αυτή την περίπτωση οι εθνικές εμπορικέ τράπεζες ε, de facto λειτουργούν ως φραγμοί. Δηλαδή αγοράζουν τα κρατικά ομόλογα. Και αυτό δημιουργεί μια στενή σχέση ανάμεσα στον κίνδυνο πτώχευση του Κράτου και κίνδυνο ε, μετατροπή του χρέου μέσω τη ε, ρευστότητα των τραπεζών. Πολύ απλά δηλαδή, εάν οι τράπεζες σε μια χώρα έχουν μεγάλο τμήμα του χρέους, το οποίο και υπάρχει δηλαδή κάποια πίεση γιατί πέφτουν όλοι πάνω για να πάρουν τα λεφτά τους πίσω, τότε ε, τα λεφτά για των, ε, των εγγυήσεων ε, μειώνονται και στην πλευρά του παθητικού των τραπεζών υπάρχει πάλι κίνδυνος να πέσουν πάρα πολλοί καταθέτες ας πούμε και να ζητήσουν τα λεφτά τους πίσω. Αυτό λοιπόν μπορεί να δρομολογήσει μια αναγκαστική έξοδο από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ευρωζώνη τέλο πάντων. Επομένω, ο κίνδυνο πτώχευση ενό κράτου ε, συνδέεται στενά με, την, ε, με τον κίνδυνο ε, μετατροπή του χρέου. Ε, η πρόταση τη Κομισιόν σε αυτό το πλαίσιο είναι μείωση του κινδύνου, ε, να έχουμε τα ασφαλή λεγόμενα στοιχεία ενεργητικού. Η πρότασή μα πάει πιο πέρα. Είναι να χωρίσουμε τον πιστοτικό κίνδυνο από τον κίνδυνο ε, μετατροπή του χρέου μέσω ε, διαφοροποίηση ε, τη έκθεση του χρέου των κρατών, ούτω ώστε να υπάρχει εξασφάλιση των εγγύσεων σε περίπτωση κρίση. Δηλαδή, οι τράπεζε πάντα να έχουν αρκετέ εγγύσει για να εξασφαλίσουν ρευστότητα από την Κεντρική Τράπεζα. Επίση, να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα εγγύηση των καταθέσεων, το οποίο θα υπάρχει πριν εμφανιστεί το πρόβλημα των ε, τοξικών δανείων, μάλλον πριν λυθεί το πρόβλημα των τοξικών δανείων. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αυτή τη στιγμή υπάρχει πιθανότητα ως τελευταία καταφυγή να αναδιαρθρώσουμε το κρατικό χρέος, το δημόσιο χρέος, τότε ο MT, δηλαδή η ΕΚΤ, μπορεί να εξασφαλίσει τον υπόλοιπο κίνδυνο, που είναι ο κίνδυνος μετατροπής του χρέους. Δεν υπάρχει δηλαδή σε καμία περίπτωση παραβίαση της συνθήκης. Το να καταστήσουμε την αναδιάρθρωση του χρέους ως τελευταία λύση, ε, να μην γίνεται αυτόματα με στην Ευρωζώνη, να είναι δυνατότητα αλλά να μην γίνεται αυτόματα. Έτσι. Αλλά θα καταστήσει την Ευρωζώνη πιο ανθεκτική γιατί θα επιτρέψει στην ΕΚΤ, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να παίξει το ρόλο της. να κρατήσει ακέραια την Ευρωζώνη με σεβασμό των συνθήκων. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας έχουμε καλέσει εσάς προσωπικά, όχι ως εκπρόσωπο κάποιου άλλου. καθηγητής Φεντερίκο Φαμπρίνη είναι ο επόμενος ομιλητής, καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου από το Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου, School of, School of Law and Government. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Uh, Χαίρομαι που είμαι εδώ στο σπίτι των Ευρωπαίων πολιτών. Θα σας μιλήσω για την αστυνομική ικανότητα ε, από συνταγματικής πλευράς και σύντομα θα ήθελα να σας δώσω την νομική ε, οπτική γωνία αυτού του νέου δημοσιονομικού εργαλείου μέσα στο κοινοτικό πλαίσιο και για την Ευρωζώνη με καθηγητής νομικής και θα συμπληρώσω αυτά που είπε η Ανιέσα που μίλησε ως οικονομολόγος και νομίζω ότι αυτά που είπε επιχειρηματολογούν υπέρ μιας ισχυρή δημοσιονομικής ικανότητας. Θα προσπαθήσω με τη δική μου ε, συμβολή να ενισχύσω τα επιχειρήματα αυτά. Η παρουσίασή μου διαρθρώνεται ως εξή. Πρώτον, θα σας παρουσιάσω τις κατεμές ταγματικές βάσεις για την ανάπτυξη μιας δημοσιονομικής καλότητας στην Ευρωζώνη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά δεύτερον, θα εξηγήσω πάλι κατεμέ ποιες είναι οι σταγματικές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αν θέλουμε να έχουμε αυτή τη δημοσιονομική ικανότητα και να είναι και επιτυχής και τρίτο. Θα προσπαθήσω να καταλήξω με κάποια αισιόδοξη νότα για αυτά που κάτε με πάντα είναι κάποιες σταγματικές ευκαιρίες για τα επόμενα έτη, τους επόμενους μήνες. Πρώτο σημείο λοιπόν, συνταγματικές βάσεις, δυνάμει ε, νομικές βάσεις. Έχω γράψει και στο δικό μου σύγγραμμα ότι υπάρχει ε, στέρεο, υπάρχουν στέρεα νομικά θεμέλια για τη μουσουλμική ικανότητα. Έχουμε το άρθρο 311 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι η Ένωση θα διαθέτει τα απαραίτητα μέσα που θα τι επιτρέψουν να φέρει σε πέρα τι πολιτικέ τη με την επιφύλαξη των εσόδων, άλλων εσόδων. Μάλλον θα χρηματοδοτείται από του ίδιου πόρου αυτό ο περιβολισμό. Αυτό το βλέπουμε σε συνδυασμό και με το άρθρο 113 της συνθήκε για τη λειτουργία Ευρωπαϊκή Ένωση που στηρίζει και αυτό την ανάπτυξη των ε, ίδιων πόρων που ασύζονται στα φορολογικά έσοδα. Αν μιλάμε τώρα συγκεκριμένα για την Ευρωζώνη και να προεπολογισμό για την Ευρωζώνη, υπάρχουν και άλλες διατάξεις ε, στις συνθήκες που θα μπορούσαν ε, να αιτιολογήσουν ε, την ανάπτυξη αυτού του νέου δημοσιονομικού εργαλείου και συγκεκριμένα το άρθρο 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δημιουργήσει μια οικονομική και νομισματική ένωση. Νομίζω ότι όταν λέμε οικονομική και νομισματική ένωση <coughs> αυτό περιλαμβάνει μια δημοσιονομική διάσταση μετά τη συνδέκη της Λισαβόνας υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα άρθρα όπως ε, και το 136 άρθρο της ε, Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τη θεσμοθέτηση της Ευρωζώνης ως ε, ένα υποσύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως δικηγόρος με ειδίκευση στα ευρωπαϊκά θέματα η δομή και το πνεύμα των συνθήκων θεωρείται αποτελεί επίσης βάση για την ανάπτυξη ενός ε, με την Ευρωζώνη. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειε, φαντάζομαι ότι θα μπορούσαμε να τα συστήσουμε στον κύριο ερωτοπαντήσεων. Η αρχή τη δημοκρατία, η αρχή της, ε, ε, του ομόσπαντου χαρακτήρα ή τη αναλυκότητα, 10 ε, και 5 άρθρα, αυτά νομίζω δικαιολογούν την ανάπτυξη αυτού του νέου μέσου, αυτού του νέου μηχανισμού στο συνταγματικό δίκαιο, όταν μιλάμε για αντιπροσώπευση, περιλαμβάνουμε την ε, φορολόγηση. Δεν μπορεί να υπάρχει, αν δεν υπάρχει αντιπροσώπευση, ε, φορολόγηση και τούμπαλιν. Και στις συνθήκες υπάρχει και η διάκριση εξουσιών και αρμοδιότητων μεταξύ ένωση και κρατών. Άρα η ανάπτυξη δημοσιονομική ικανότητας είναι κάτι πολύ σημαντικό αν θέλουμε να διατηρήσουμε τη διάκριση των εξουσιών. Δεν <clears throat> θα πω ότι είναι απλά νομικώς ε, εφικτή η μουσουλμική ικανότητα, αλλά θα έλεγα ότι είναι και απαραίτητη. Τώρα, η ανάπτυξη νέας δημοσιονομικής ικανότητας για την οικονομική σταθεροποίηση. Έρχεται αντιμέτωπη με σημαντικέ σταγματικές προκλήσεις. Δεν είναι απλή, ε, απλές, ε, απλή προβληματισμοί, διακοσμητική, αλλά ουσιώδη ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο σχεδιασμό αυτού του νέου μέσου. Τρεις βασικές προκλήσεις. Η πρόκληση της ασυμμετρίας, η πρόκληση της ομοφωνίας και η πρόκληση της αντιπροσώπευσης. Πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε και τις τρεις προκλήσεις αυτές. Με συντομία να σχολιάσω αυτές τις τρεις βασικές προκλήσεις. Ασυμμέτρια. Όπως γνωρίζετε, ασυμμετρία μάλλον, όπως γνωρίζετε, υπάρχει ασυμμετρία σε αυτό το μέγεθος, την οικονομική ισχύ, τον πλούτο, τη θέση στον ε, επιχειρηματικό κύκλο μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Είναι ασυμμετρικά μεταξύ τους και αυτό επηρεάζει και το δημοσιονομικό διάλογο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά τα κράτη αν είναι καθαροί εισφορείς ε, ή δικαιούχοι. Και δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα με αυτές τις μεταφορές ε, πιστώσεων τα τελευταία ε, χρόνια και μέχρι το τελευταίο δημοσιονομικό πλαίσιο. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια δημοσιονομική ικανότητα, θα πρέπει να απομακρυνθούμε από το μοντέλο που ουσιαστικά περιχαρακώνει τι ασυμμετρίε μεταξύ των κρατών μήλων ε, και βασίζεται για τη χρηματοδότηση στις μεταφορές πιστώσεων, αλλά θα μεταφερθεί, θα αλλάξει και θα γίνει ένα νέο σύστημα. Η δημοσιονομική ικανότητα θα χρηματοδοτείται από γνήσιους ίδιους πόρους που θα παράγονται λόγω ακριβώς της ύπαρξης της ίδιας της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν δεν σπάσουμε το φαύλο κύκλο αυτών των διακρατικών εμβασμάτων των πιστώσεων κινδυνεύουμε η δημοσιονομική ικανότητα να υποστεί ε, πλήγματα από αυτή τη δυναμική που ξέρει πολύ καλά και ο κύριος Ρέγκλινγκ από τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και με ανησυχεί κάπω η ιδέα ότι θα μπορούσαμε με την απλή κοινοτικοποίηση, η συμπερίληψη του ESM στη, στο κοινοτικό κεκτημένο να έχουμε ακριβώ αυτή τη δημοσιονομική ικανότητα. Παναλαμβάνω, θέλουμε γνήσιου ίδιου πόρου για τη χρηματοδότηση του προεπιλισμού τη Ευρωζώνη. Και εδώ έχουμε μια διαφορετική πρόκληση να αντιμετωπίσουμε που θα την έλεγα πρόκληση της ομοφωνίας. Στην, ε, στις όλα τα δημοσιονομικά, χρηματοοικονομικά ζητήματα υπόκεινται στο νόμο της ομοφωνίας που σημαίνει ότι μπορεί κάθε κράτος ε, να ε, προβάλλει βέτο. Ένα σύστημα που θα βασίσει στην ομοφωνία σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει συνένεση. Και θα είναι δύσκολο να σημειωθεί πρόοδο. Τι έχει γίνει στον τομέα αυτό. Οι συνθήκε προβλέπουν κάποια εργαλεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ελαχιστοποίηση του προβλήματο. Ενισχυμένη συνεργασία, για παράδειγμα ώστε κράτη συγκεκριμένα να μπορούν να αναλαμβάνουν δράση όταν δεν ε, υπάρχει προθυμία από το σύνολο των κρατών μελών. Όμως, ε, αν θέλουμε να είμαστε και δίκαιοι, αυτό δεν είναι το βέλτιστο δυνατό εργαλείο, διότι τα αφορολικά ζητήματα από μια δέσμη κρατών δεν ε, έχουν και πάντοτε ευτυχή κατάληξη. Από νομικής σκοπιάς λοιπόν το ζήτημα τη ομοφωνία, τη δεκαετία λήψη αποφάσεων για τα δημοσιονομικά και χρηματοοικονομικά συστήματα με ομοφωνία πρέπει να αντιμετωπιστεί και ανέκυψε και στην τελευταία συνταγματική συνέλευση. Ε, θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Τέλο, ναι, μεν προχωράμε προ την κατεύθυνση του να περκεράσουν τι προκλήσει τη ομοφωνία, αλλά προκύπτει μια άλλη ε, πρόκληση για τη δημοσιονομική ικανότητα. Είναι η πρόκληση τη αντιπροσώπευση, representation αν δεν υπάρχει αντιπροσώπευση, δεν υπάρχει φορολόγηση, όπως είπα. Αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και σε κάθε άλλο πλαίσιο. Και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο σε ό,τι αφορά την λήψη αποφάσεων για τα φορολογικά ζητήματα. Είναι απαράδεκτο από δημοκρατική πλευρά, η δημοσιονομική ικανότητα να αποφασίζεται χωρίς να έχει φωνή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να συνοψίσω λοιπόν, κατά την άποψή μου, μια επιτυχημένη δημοσιονομική ικανότητα θα πρέπει να αποφύγει ε, το ε, κακό αυτό των ε, διακρατικών μεταφορών πιστώσεων. Θα πρέπει να επεκεράσει το πρόβλημα της αρνησικυρίας, του βέτο από κάποιο κράτος και τέλος βέβαια πρέπει να ξεπεράσει τα προβλήματα της αντιπροσώπησης. Δηλαδή πρέπει να ακούγεται η φωνή των πολιτών, η φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Φιλόδοξη ε, αυτή η λίστα με τις προκλήσεις. Εγώ όμως είμαι αισιόδοξο εκφύσεως, γι' αυτό λοιπόν βλέπω και κάποια παράθυρα ευκαιρίας για το μέλλον. Ίσως να είναι ηρωνικό ε, για κάποιο περίπτωση δηλαδή, αλλά θεωρώ το Brexit δίνει, ε, μας δίνει κάποια περιθώρια ισοδοξίας, Γιατί η απόφαση αποχώρησης από, από την Ένωση για το Ηνωμένο Βασίλειο δημιουργεί μια τρύπα στη χρηματοδότηση σε ένωση για την επόμενη περίοδο, το επόμενο πολιετές. Και έτσι πρέπει να βρεθούν πόροι για τη χρηματοδότηση του προπολογισμού. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια το Κοινοβούλιο ενέκρινε δύο ψηφίσματα για του ίδιου πόρου και για το ε, μέλλον ε, του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Το επόμενο πολιτικό Πολύ φιλόδοξα τα ψηφίσματα αυτά. Και ο στόχο είναι ότι αν ε, δεν προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε πέραν του να πούμε απλά έχουμε ένα κενό, μια τρύπα στον πολεμισμό και ζητάμε χρηματοδότηση, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με άλλο τρόπο, να πείσουμε τα κράτη-μέλη να χρηματοδοτήσουν πραγματικά τη δημοσιονομική ικανότητα για την Ευρωζώνη. Επίσης, κάτι που δεν έχει συζητηθεί μέχρι στιγμή ευρέως, αλλά άπαξ και έχει αποχωρήσει από την Ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο, τα υπόλοιπα, τα αναπόμενα 27 κράτη-μέλη θα είναι υποχρεωμένα να προχωρήσουν σε μια σειρά βαθιών σταγματικών μεταρρυθμίσεων. Τη συζήτηση ε, την ξεκίνησε πρόσφατα το Κοινοβούλιο όταν ψήφισε για την σύνθεση του προσεχούς Κοινοβουλίου, την ε, κατανομή, την αναδιανομή των ευρών. Αλλά θα χρειαστούν και άλλες αλλαγές όταν το Ηνωμένο Βασίλο πάψει να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι και πάλι και αυτό είναι ένα παράθυρο ευκαιρίας για να αντιμετωπιστούν κάποια δομικά ζητήματα, όπως αυτά που σας παρουσιάσα προηγούμενη, ε, στις προηγούμενες διαφάνειες. Υπάρχουν λοιπόν λόγοι αισιοδοξία. Υπάρχουν περιθώρια για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Βέβαια, <clears throat> αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον της ΟΝΕ και την ανάπτυξη ενός προπολογισμού για την Ευρωζώνη, η οποιαδήποτε αυτή η συζήτηση θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλη συζήτηση για το μέλλον τη Ευρώπη, όπω για την Αμυντική Ένωση, για παράδειγμα. Γιατί τελικά δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το χάσμα μεταξύ των βόρειων και των νότιων χωρών, ε, όταν συζητάμε την ΟΝΕ, όλα τα κράτη-μέλη αντιλαμβάνονται τις μείζονες γεωπολιτικές προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουν. Για να τις αντιμετωπίσουμε πρέπει να έχουμε μια αμυντική ένωση που γι' αυτό απαιτείται επίσης ένας κοινό προπολογισμό. Ήμουν πολύ σύντομο και ζητώ συγγνώμη. Αλλά ως ακαδημαϊκός να μην διαφημίσω κι εγώ το έργο μου. Έχω συγγράψει ένα βιβλίο για την οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη και ένα άλλο για το Brexit. Έτσι για να έχετε περισσότερη βιβλιογραφία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε καθητά. Τώρα, ο Χόρχε Νούνιας από το Κέντρο Ευρωπαϊκών ε, Μελετών Πολιτικής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που με φιλοξενείτε εδώ. Ε, εξέτασα αυτό το θέμα έχοντας κατά νου τη σταθεροποίηση, ιδιαίτερα τη σταθερότητα και ποιο είναι ο ρόλος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Θα ξεκινήσω ε, και θα πάω κάπου αλλού, θα το δω από άλλη οπτική ε, γωνία και θα επανέλθω μετά στον προπολογισμό. Γιατί έχω εξετάσει άλλα θέματα. Ε, ε, εσείς μπορείτε να δείτε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και να βρείτε λύσεις εκεί, αλλά έχω βρει μεγάλο δυναμικό στους εθνικούς λογαριασμούς των κρατών μελών και έχω ε, μελετήσει αυτό το θέμα. Αυτό θα ήθελα να πω ότι είναι η δημοσιονομική ικανότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, πρέπει να δούμε ε, τι, τι αντιδραστικά μέσα μπορούμε να βρούμε, αλλά θα πρέπει να δούμε και τι προληπτικές ικανότητες, πώς να προλάβουμε, πώς να μετριάσουμε τα προβλήματα και τις κρίσεις του μέλλοντος και νομίζω δεν έχει μελετηθεί επαρκώς και να μην δημιουργήσουμε κάτι που να αντιδρά απλώ αλλά κάτι που να μας προλαβαίνει από αυτό τον αντίκτυπο των κρίσεων. Ε, άρα δεν νομίζω ότι έχουν αντιμετωπιστεί τα αίτια από την εξάδα των μέτρων. Θα ήθελα να πω ότι δουλεύω μια ομάδα ατόμων από τη ΣΥΠΑ, από τη Νέα Ζηλανδία και είναι ειδική και εξετάζουμε την αξία και την σημασία της δημοσιονομικής διαχείρισης και την σταθερότητα. Και σε σχέση, ε, δυστυχώς, ε, τα κράτη-μέλη ε, δεν το διαχείριζονται σωστά. Άρα υπάρχουν και σύμφωνα με την ομάδα μας βλέπουμε βλέπουμε ένα πόλης του ΑΕΠ διαχρονικά και υπάρχει ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ μέσα από τους μηχανισμούς συντονισμού αλλά αυτό έχει αποκλειστεί από πολλά κράτη-μέλη. Αυτό το κατανοούν και ο και το Ευνουτού και αρχίζουν να λένε κοιτάξτε το αυτό το θέμα, αλλά ε, τελικά ανετίθεται συζήτηση σε λογιστές και το έχουμε εξετάσει αυτό το θέμα με την ομάδα, αλλά έχω συνειδητοποιήσει ότι είναι σημαντικό και παραμένω σε αυτή την ομάδα και το εξετάζουμε εδώ και πάνω από χρόνο. Ε, σημαίνει ότι υπάρχει μια υποκείμενη αδυναμία να ελέγχουν τους, ε, τις ίδιες τις κυβερνήσεις. Το είδαμε στην Ελλάδα όπου ανακάλυψαν ότι υπήρχε ε, διονκωμένο πρόβλημα που δεν είχε αναφερθεί. Θα πρέπει να αποφεύγεται αυτό διότι επηρεάζει την πιστοληπτική ικανότητα και αυξάνει το σοκ. Υπάρχουν τρόποι επίλυσης και λέω ότι υπάρχει ε, θα πρέπει να γίνει όχι μόνο μεταρρύθμιση του προπολογισμού, κάτι άλλο. Η ομάδα αυτή το εξετάζει, εξετάζει ε, τα πρότυπα των δημόσιων ε, λογαριασμών, των ε, διεθνών λογιστικών προτύπων και βλέπουμε ποια είναι η, ε, ποια είναι η αξία των στοιχείων των περιουσιακών στοιχείων. Θα πρέπει έχω στην Πορτογαλία είναι η πρώτη χώρα που έχει πλήρη μεταρρύθμιση σε όλα τα συστήματα δημοσίων ε, λογαριασμών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και το κάνουν διότι συνειδητοποίησαν ότι μπήκαν τόσο βαθιά που δεν ήξεραν ποια ήταν τα περιουσιακά στοιχεία, πολλά πράγματα που επηρέαζαν την πιστοληπτική ικανότητα και αυτό τους βοηθάει πολύ. Πρώτα απ' όλα, ε, η σταθερότητα ξεκινάει με καλή διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στήριξη της σταθερότητας από τη βάση. Να πούμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν 50% της οικονομίας στα χέρια τους, ανάλογα με τη χώρα, κατά μέσο όρο 46%, πριν από μερικά χρόνια τώρα, από το 2015 είναι αυτός ο πίνακας και μέχρι και 58%. Είναι πολλά χρήματα ε, στα χέρια της κάθε χώρας και υπολογίζεται 45 ε, εκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Ε, μόνο ε, σε 15 ε, Υπάρχει πρόβλημα λήψη αποφάσεων και πρέπει να πω ότι υπάρχουν αυτά τα πράγματα που έχω σβήσει. Μερικές χώρες δεν αναφέρουν τις υποχρεώσεις σε συντάξεις. Δεν έχουμε κανονικά πρότυπα. Δεν βλέπουμε ποια είναι η σταθερότητα της χώρας όταν την πλήττει ένα σοκ. Θα επανέλθω στο προπολογισμό, αλλά πιστεύω αυτό είναι τόσο σημαντικό και το έχουμε παραβλέψει τόσο πολύ όταν με ρωτούν τι μπορεί να κάνει ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση όταν υπάρχει κρίση. Λέω, δεν είναι καλύτερα να δούμε τι μπορεί η χώρα να κάνει και μετά να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Λοιπόν, ε, η κυβερνήσεις πολλές φορές δεν χρησιμοποιούν τα βασικά εργαλεία διαχείρισης. Ε, αντί να βλέπουν τον ετήσιο προϋπολογισμό, να βλέπουν την μακροπρόθεσμη σταθερότητα και να βλέπουν την κυκλική συμπεριφορά. Πρέπει να βλέπεις κάθε φορά τις επενδύσεις εξίσου ετησίω. Ας δούμε τώρα τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και τη σταθεροποίηση. Ο, αυτό, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα πρέπει να έχει ρόλο στη σταθεροποίηση. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μακροοικονομική σταθεροποίηση. Είναι μικρός ο προϋπολογισμός και είναι σχεδιασμένος ως εργαλείο επένδυσης. Θα πρέπει να επανεφευρεθεί, θα πρέπει να δούμε τις άμεσες πληρωμές ε, στη γεωργία, η ανακατανομή, τη συζητάμε 30 χρόνια δεν το έχουμε επιλύσει και πολλές φορές έχουμε συζητήσει τεράστιες μεταρρυθμίσεις του προπολογισμού και έχει πάρει τόσο χρόνο για τις αμέσες πληρωμές και αναρωτιέμαι πώς θα επιληθεί. Μπορεί να φαίνομαι ή να ακούγομαι ότι δεν είμαι και πολύ θετικός, αλλά ε, αναρωτιέμαι μετά από τόσα χρόνια. Είναι άκαμπτος ο προπολογισμό, είναι αδρανής, έχει περιορισμένα εργαλεία, έχει το Ταμείο Αλληλεγγύης, το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων. Αυτή η πρωτοβουλία έχει μεταφέρει ε, ε, δεν έχει αυξήσει όμω τον προπολογισμό. Αν πρέπει να μεταφερθούν κονδύλια και αν, υπάρχει κρίση το 2019, τι θα γίνει, θα πάρουμε τα χρήματα του μέλλοντος που δεν υπάρχουν, διότι δεν μπορεί να μετατοπίζονται κονδύλια ε, από, το, από παρελθόν στο μέλλον. Δεν έχει σημασία πόση ευελιξία, αλλά δεν έχεις, δεν έχεις όμως τα κονδύλια. Αυτά είναι πράγματα που δεν τα έχουμε μελετήσει, δεν έχουν μελετηθεί και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Το τρίτο μάθημα είναι ότι ο ευρωπαϊκός προπολογισμός μπορεί να εκτελέσει κάποιες, κάποια περιορισμένη οικονομική σταθεροποίηση. Ναι, μπορούμε να ξεκινήσουμε, ε, αλλά να μην ε, υποσχόμαστε πολλά που να μην ε, τα τηρήσουμε στο τέλος. Έχουμε την περιοχή, την Σέγγεν, έχουμε τους γεωργικούς τομείς, άλλους τομείς και όταν υπάρχει μια κρίση δεν υπάρχουν τα κονδύλια, μεγάλο το σοκ. Είναι καλύτερο να αποφύγουμε τώρα κάποιο κονδύλι που να μην είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το σοκ. Τι μπορεί να κάνει ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός. Όταν δείτε τα μακροοικονομικά, έχουμε, δύο, έχουμε την το σκεπτικό, τα εργαλεία πολιτικής και τα κυριότερα στοιχεία. Έχουμε την μακροχρηματοπιστική σταθερότητα και την οικονομική σταθερότητα. Το θέμα είναι, αυτά τα, το ESM θα πρέπει να είναι εκτός όταν ε, μιλάμε για στήριξη του συζυγίου πληρωμών και σοκ και θα εξηγήσω γιατί σε λίγο. Και υπάρχει οικονομική σταθεροποίηση, ο προπολογισμό μπορεί να έχει σχέση, αλλά υπάρχουν ε, θέματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Και θα είναι δύσκολο, διότι αλλάζει στη φύση του προπολογισμού και απαιτεί τι σωστές δομές. Τι ρόλο μπορεί να παίξει λοιπόν ο προπολογισμό. Έχουμε το πιο εφικτό στόχο να ενισχύσουμε τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, τα ΕΔΕΤ, να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν εκεί επενδύσεις για να δημιουργηθεί, να ανθεκτικότητα, ε, να μην υπάρχει τόση απορρόφηση, να δημιουργηθεί περαιτέρω μελλοντική αξία. Υπάρχουν θέματα που ήδη ξεκίνησαν, πολλά έχουν γίνει, πολλά μπορούν να γίνουν ακόμη και μπορεί να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, δεν θα, με κάποιες συμφωνώ, με κάποιες άλλες, με κάποιες όχι. Έχουμε και ένα έγγραφο περισυλλογής για την το Ευρωπαϊκό Σύστημα Προστασίας των Επενδύσεων, για το Ταμείο για τις Δύσκολες Μέρες, αλλά αυτό το έγγραφο δεν αναφέρεται συγκεκριμένα, ε, δεν βλέπω το ένα να αντανακλά το άλλο ε, τα, έγγραφα της, της Επιτροπής. Θα πρέπει να σκεφτούμε τι ακριβώς ε, παρουσιάζουμε. Θα πρέπει Αυτά είναι τα διαρθρωτικά ταμεία ε, και ίσως να υπάρχει και αυτό το ταμείο για τις δύσκολες μέρες. Να δημιουργήσουμε αυτό τον ε, χρηματοπιστωτικό χώρο για να το κάνουμε αυτό μέσα στο προπολογισμό. Πρέπει να υπάρχει όμως η δυνατότητα και αυτό θα είναι δύσκολο με το 1%. Τελευταία διαφάνεια, το σχέδιο προστασίας των επενδύσεων, για να αποφευθεί η κάμψη των επενδύσεων, τι σύσταση πρέπει να έχει, με ποια εργαλεία, με ποια μέσα, ποιες προβλέψεις. Το θέμα είναι ότι είμαστε, θα έχουμε την πρόταση για το MFF πολύ σύντομα. Πώς, σε ποιο βάθμο μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτά τα υπέροχα σχέδια, θα προταθεί, όχι, δεν ξέρω. Το σύστημα αντασφάλισης για την ανεργία, είναι διαφορετικά τα συστήματα στα κράτη-μέλη. Πώς μπορούμε να το κάνουμε με σαφήνεια, ακούσαμε. Και ίσως να αληθεύει ότι δεν θα πρέπει να περιέχεται στο προπολογισμό ή το Ταμείο Εκτάκτων Περιστατικών. Θα ήταν καλό να είναι αντιδραστικό και γρήγορο, αλλά πόσο μεγάλο. Τι γίνεται όταν δεν υπάρχει; ε, Δεν μπορεί, όταν δεν μπορεί λοιπόν, πια να δανειστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ερωτηματικά που παραμένουν ανοιχτά και όταν είναι περιορισμένο ο προπολογισμό, θα πρέπει να αναρωτηθούμε πώ θα κάνουμε εκτό και να αυξηθεί ο προπολογισμό σε μεγάλο βαθμό. Και δεν το ακούμε αυτό ούτε από την ε, ε Κομισιόν ε, και ξέρουμε γιατί. Ο προπολογισμό τη Ευρωζώνη επίση υπάρχει μια ερώτηση ίσως ε, να μην ήταν κακό τα κράτη-μέλη να εξετάσουν αυτά τα πράγματα. Ε, δεν ξέρω όμως αν πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος προπολογισμό. Ε, αν γίνει, θα μπορούσε να γίνει με την αύξηση του ευρωπαϊκού προπολογισμού και να καλυφθούν οι χώρες εκτός της Ευρωζώνης. Γιατί όταν γίνει το Brexit, αν αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτοί που δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης ίσως να υπάρχει τρόπος να βοηθηθούν ή να ενταχθεί το, το ισοζύγιο πληρωμών τους μέσα στο σύστημα της Ευρωζώνης για να έχουν τη στήριξη από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Σημαίνει ότι θα γίνει κάποια μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού σε μεγάλο βαθμό. Δεν θα τα δω όλα τα σημεία, αλλά τι κάνουμε με το 1%. Το μεγάλο ερώτημα, το 1% θα παραμείνει. Την περασμένη εβδομάδα ε, ήμουνα σε μια συνάντηση υπουργών οικονομικών και ήταν ε, σαν να μιλούσαμε κινέζικα. Ε, με ενόχλησε αυτό, αλλά είναι πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, ε, for this note. Ευχαριστώ. Και για αυτό το τελευταίο που είπατε, που είναι ρεαλιστικό. Ξέρουμε πολύ καλά ποιο είναι το πολιτικό μας περιβάλλον. Ξέρουμε ποιες είναι οι θέσεις των κρατών μελών. Είναι δύσκολο να παντρέψουμε τους διάφορους στόχους. Και επομένως νομίζω είναι και η ώρα να ακούσουμε και την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ τον ε, εκπρόσωπο της ΕΚΦΗΝ που ήρθε εδώ για να μας ε, παρουσιάσει τη θέση της ε, Κομισιόν και για την ΟΝΕ και για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ξέρουμε το πακέτο ποιο είναι, ξέρουμε τους περιορισμούς και πέρα από τα σχόλια που θα πρέπει να κάνετε για αυτά που ακούσατε, θέλουμε να ακούσουμε και εμείς τι μας περιμένει. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε για να σχολιάσουμε Καλωσορίζουμε αυτή την εκδήλωση. Είναι μια πρωτοβουλία που είναι απόλυτη σημασία, υψίστη σημασία για μα, προκειμένου να μην ανοιχτή συζήτηση για το θέμα αυτό. Ειδικά το θέμα τη λειτουργία τη δημοσιονομική σταθερότητα που θεωρούμε είναι εκ των όνου κάνευ για την ολοκλήρωση, για την ολοκλήρωση τη ΟΝΕ. Αυτή η συζήτηση δεν γίνεται εν κενό. Έχουν γίνει έχουν ετοιμαστεί πολλές εκθέσεις πρόσφατα τα τελευταία χρόνια που ζήτησαν τη δημιουργία ε, δημοσιονομικής ικανότητας στην Ευρωζώνη και κυρίως ε, μιας ε, λειτουργίας δημοσιονομικής σταθεροποίησης. Υπήρχε η έκθεση των τεσσάρων προέδρων ε, το 2012 υπό την αιγύδα του Φαντεν Πόι και η έκθεση των πέντε προέδρων το 2015 υπό την αιγύδα του πρόεδρου Γιούνκερ. Ε, το έγγραφο προβληματισμού της Κομισιόν που δημοσιεύθηκε πέρυσι το Μάιο και τέλος και σημαντικό το ψήφισμα που υιοθετήθηκε από το Κοινοβούλιο στις 16 Φεβρουαρίου του 2017 με βάση την έκθεση Μπέγκε και Περές. Και ακόμα πιο πρόσφατα ακούσατε από την ΕΚΤ, το Δουνουτού, τον ΩΣΑ πολλά επιχειρήματα υπέρ της δημιουργίας μιας, ενός μηχανισμού δημοσιονομικής ε, σταθεροποίησης. Ό,τι αφορά το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζήτησε τη δημιουργία αυτής της δημοσιονομικής ικανότητας επιπροσθέτως και χωρίς ε, να δημιουργείται πρόβλημα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό σταθερότητα. Η δημοσιονομική ικανότητα με βάση αυτό το ψήφισμα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει ένα κώδικα σύγκληση που θα εστιάζει στην φορολογία, στην αγορά εργασία, στι επενδύσεις, στην παραγωγικότητα, κοινωνική συνοχή, καλή διακυβέρνηση. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ικανός απορρόφησης των ασύμετρων σοκ και θα πρέπει να είναι ουδέτερο συν το χρόνο για να μην έχουμε μόνιμες μεταφορές ε, πιστώσεων. Και το τρίτο στοιχείο του ψηφίσματος είναι ότι θα πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίζει τα συμμετρικά σοκ, τα οποία επηρεάζουν πολλαπλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτόχρονα. Επιπροσθέτως, όπως υπόθηκε και στην αρχή, ε, το ψήφισμα ζητούσε την ανάπτυξη ε, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και το μηχανισμ τη μετατροπή του σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Υπάρχει λοιπόν ε, ευρεία, αν όχι ομοφωνία, υπάρχει ομόφωνη, συγγνώμη, συνένε, ε, αυξημένη συνένεση ότι η Ευρωζώνη χρειάζεται ένα κεντρικό μηχανισμό σταθεροποίησης, δημοσιονομικής σταθεροποίησης. Ας σας εξηγήσω γιατί πιστεύουμε ότι είναι βασικό για την Ευρωζώνη αυτό. Πριν ε, μπω πολύ γρήγορα στα στοιχεία τα οποία βάλαμε εμείς επιτάπητος το Δεκέμβριο. Η Ευρωζώνη αντιμετωπίζει πολύ, ε, μια πολύ, έχει μια πολύ συγκεκριμένη δομή. Η ενιαία νομισματική πολιτική αφορά το συνολικό επίπεδο, έτσι, τις συνολικές διακοιμάσεις, ενώ η δημοσιονομική πολιτική είναι αποκεντρωμένη και καταρχήν μπορεί να ανταποκριθεί μόνο στα ειδικά σοκ που αντιμετωπίζουν οι επιμέρους χώρες μέσω της ε, του Εθνικού Μηχανισμού Δημοσιονομικής Σταθεροποίησης. Αυτό λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες και λειτουργεί καλά, αλλά είναι ανεπαρκές όταν υπάρχουν σημαντικά μακροοικονομικά σοκ, όπως αυτά που είδαμε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης. Σε περιπτώσεις τέτοιου τύπου, ε, η εθνική δυνατότητα δημοσιονομικής σταθεροποίησης τρίβεται ε, λόγω της πίεσης της αγοράς περιορίζεται, αντιμετωπίζει πιέσεις και ακόμα και τα κράτη που έχουν ε, ε, υγιή δημοσιονομική θέση, όπως ας πούμε η Ιρλανδία και η Ισπανία το 2008 όταν τσέπληξε η κρίση, είχαν μια δημοσιονομική κατάσταση που ήταν σύμμορφη προς τους κανόνες και παρόλα αυτά ας πούμε όταν αντιμετώπισαν αυτό το σοκ που έγινε το 2010 και 2011, μπορεί να θυμάστε ότι διάφορα κράτη-μέλη κατέρευσαν κατέρευσαν τα έσοδά τους και φτάσαν σε επίπεδα 2% του ΕΠ ανάμεσα στο 2010 και το 2011. Και αυτό οδήγησε σε ουσιαστική επιδείνωση των δημοσιονομικών ελλημάτων και σε ορισμένε περιπτώσεις σε αυτές τις προβληματικές χώρες είχαμε φτάσει στο μείον 16% του ΑΕΠ. Δηλαδή, ε, ο μέσος όρος ε, στην Ευρωζώνη το 2010 ήταν μείον 6% του ΑΕΠ, των δημοσιονομικών ελλημάτων παντενό. Ένα τρομακτικό δημοσιονομικό σοκ. Όταν λοιπόν υπάρχει και πίεση της αγοράς, η οποία ακολουθεί, περισσότερες χώρες μπαίνουν σε μια γρήγορη διαδικασία εξυγίανσης. Και αυτό οδήγησε σε προληπτικές, ε, προκυκλικές συγγνώμη, δημοσιονομικές πολιτικές. Αυτό είδαμε να γίνεται στην Ευρωζώνη το 2011 και μέχρι το 2015 μία περίοδο όπου η δημοσιονομική θέση της Ευρωζώνης συνολικά ε, περιορίστηκε σε μία εποχή όπου το κενό με την παραγωγή ας πούμε ε, ήταν ουσιαστικά αρνητικό. Αυτό επηρέασε και την παραγωγή, το παραγωγικό δυναμικό και έγινε και απόλυτη θέση εργασία ε, λόγω των σοκ. Αυτό είναι ένας από τους βασικούς λόγους για την πολύ ελαφρά έτσι, χλιαρή ανάκαμψη της Ευρωζώνης μέχρι πέρυσι, ειδικά όταν την συγκρίνουμε με τις ΗΠΑ και πώς αντέδρασαν μετά την κρίση. Οι ΗΠΑ ανέκτησαν τα επίπεδα πρώτης κρίσης, ε, την παραγωγή δηλαδή πρώτης κρίσης το 2011, ενώ εμείς χρειαστήκαμε στην Ευρωζώνη τέσσερα επιπλέον χρόνια για να φτάσουμε στα επίπεδα παραγωγής πρώτης κρίσης. Φτάσαμε δηλαδή μέχρι το 2015 για να ανακτήσουμε το επίπεδο προκρίσης. Η έλλειψη ενός ε, κεντρικού μηχανισμού δημοσιονομικής ε, σταθεροποίησης ε, βαρύνει πολύ την ΕΚΤ και είναι υποχρεωμένη να πάρει έκτακτα μέτρα για να παίξει το με βάση τις αρμοδιότητές της. Η ατελής αρχιτεκτονική δομή της Ευρωζώνης θεωρείται από τους επενδυτές ως βασική πηγή κινδύνου διάλυσης, δηλαδή κίνδυνος ε, μετατροπής του χρέους εννοείται εδώ. Αυτός ο κίνδυνος έγινε πολύ ορατός κατά τη διάρκεια της κρίσης και ανάγκασε την ΕΚΤ να αναγγείλει το OMT, τον, τις μόνιμες, το OMT, τις μόνιμες ε, νομισματικές συναλλαγές. Ε, αυτό εξηγεί τις, τη φτωχ... τις κακές μας επιδόσεις σε σχέση με, την, με τη ΣΥΠΑ και λόγω της απουσίας της ε, Τραπεζικής Ένωσης και της Κεφαλαϊκής Ένωσης. Και σε αυτά τα επίπεδα κάνουμε πρόοδο, αλλά πολύ αργά. Έχουμε ε, ενοποιημένη τραπεζική εποπτεία τώρα και μηχανισμό εξυγίασης των τραπεζών, αλλά δεν υπήρξε πρόοδος ε, στις συζητήσεις για το ενιαίο σύστημα εγγύηση των καταθέσεων και για τη δημιουργία ενός μηχανισμού στήριξης του του ενιαίου Ταμείου Ξεξυγίανση. Και αυτά είναι προβλήματα. Το να έχουμε μια πλήρη τραπεζική ένωση θα βελτιώσει πάρα πολύ την, τη διασπορά του κινδύνου με τον ιδιωτικό τομέα, αλλά μην πιστέψετε ποτέ ότι αυτό αρκεί, αυτή η διασπορά του κινδύνου. Φυσικά υπάρχουν στοιχεία ότι η διασπορά του κινδύνου και ο επιμερισμός με, ε, με τον ιδιωτικό τομέα ε, θα μας οδηγήσει σε κυκλικές πολιτικές. Ε, η δυνατότητα ε, σταθεροποίησης του είναι πολύ αδύναμη. Ακριβώς λοιπόν σε αυτές τις εποχές μεγάλων κινδύνων ε, μία λειτουργία σταθεροποίησης είναι απαραίτητη γιατί ο ιδιωτικός τομέας θα πάρει μέρος του κινδύνου αλλά πιο αποτελεσματικά μόνο όταν συνεργαστεί και υποστηριχθεί από τον δημόσιο τομέα και όταν υπάρξει διασπορά του κινδύνου ανάμεσα στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Φυσικά, μια κεντρική λειτουργία σταθεροποίηση δεν θα πρέπει να είναι ο πρώτο μηχανισμό άμυνα. Ο πρώτο μηχανισμό άμυνα θα πρέπει να είναι ε, μια εύρυθμη κεφαλαιακή αγορά. Αυτή, αυτό εξασφαλίζει ότι η απορρόφηση των σοκ και ο επιμερισμός ε, του κινδύνου ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα λειτουργεί καλά. Γι' αυτό πρέπει να ολοκληρώσουμε την ε, Τραπεζική Ένωση και Κεφαλαϊκή Ένωση. Επίση, το δεύτερο είναι η χρηστή δημοσιονομική πολιτική που εξασφαλίζει την οικοδόμηση ε, δημοσιονομικών ε, αναχωμάτων σε δύσκολε στιγμέ και εξασφαλίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα σοκ. Η τρίτη γραμμή άμυνα είναι η λειτουργία αυτή σταθεροποίηση. Πριν φτάσουμε στην τελευταία γραμμή άμυνας, που είναι ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμός σταθερότητα σε περίπτωση που έχουμε ε, απώλεια της πρόσβασης στις αγορές. Αγορές. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η κοινή λειτουργία σταθεροποίηση δεν είναι αποτελεσματικό εργαλείο για τον επιμερισμό του κίνδυνου, αλλά είναι σημαντικό για να μειωθούν οι κίνδυνοι για όλη τη ζώνη. Με βάση την εμπειρία των προγραμμάτων, η μείωση της πιθανότητας ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας ή ενός μελλοντικού ευρωπαϊκού νομισματικού ταμείου είναι τεράστιο όφελος και για τις χώρες που δανείζουν και για τις χώρες που δανείζονται. Ποιε είναι οι βασικές αρχές λοιπόν αυτής της λειτουργίας σταθεροποίησης. Πολύ σύντομα. Δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μόνιμες ε, μεταφορές πιστώσεων, θα πρέπει να μειώσει τον ηθικό κίνδυνο, να μην ε, επικαλύψει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας κάθετο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο θα πρέπει να αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου, θα πρέπει να είναι ανοιχτό σε μέλη που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη. Πρόσβαση στην ε, σταθεροποίηση θα πρέπει να γίνεται αυστηρά υπό όρους, με σαφή κριτήρια και ισχυρές και καλές και υγιείς πολιτικές. Τέλος, θα πρέπει να υποστηρίζει τη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες πραγματι... στην πραγματικότητα η λειτουργία αυτής της σταθεροποίησης μπορεί να στηθεί με ένα τέτοιο τρόπο που ενισχύει την συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Ε, τώρα, μετά σας κάνω μια μικρή επισκόπηση για το τι παρουσιάσαμε το Δεκέμβριο ε, σε αυτό το πακέτο που παρουσιάσαμε τότε. Μεταξύ άλλων, να σας παρακαλέσω λιγάκι να το επιδείξετε αυτό, γιατί το ξέρουμε αυτό το πακέτο, έτσι. Μας ενδιαφέρει το βασικό πακέτο, όχι του Δεκεμβρίου αν μου επιτρέπετε, ε, για να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τον λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Εντάξει. Εγώ απλά θα σας δώσω μία προεπισκόπηση του τι έρχεται στη συνέχεια. Καταθέσαμε λοιπόν επιτάπητος ιδέες για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτή η σταθεροποίηση. Τρεις συνιστώσεις. Μία γραμμή ρευστότητας από το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο που θα μπορούσε να παρέχει δάνεια τα οποία ε, θα τα εγγυάται ο ευρωπαϊκό προπολογισμό. Ένα δεύτερο συστατικό, μια δεύτερη συνιστόσα θα μπορούσε να είναι υποστήριξη από τον νοσιακό προπολογισμό και η τρίτη συνιστόσα θα μπορούσε να είναι ένα ασφαλιστικό μηχανισμό ε, με εθελοντικέ εισφορέ από τα κράτη-μέλη. Αυτή η τρίτη συνιστόσα θα μπορούσε στον χρόνο να δημιουργηθεί για να έχετε μια εικόνα πώς βλέπουμε τα πράγματα ποια θα ήταν τώρα τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα κριτήρια ενεργοποίησης. Όπως είπα, η πρόσβαση στη λειτουργία σταθεροποίησης ε, θα πρέπει να διέπεται από αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις. Άρα και αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητας πρέπει να ισχύουν. Όποιοι τηρούν το εποπτικό πλαίσιο, όποια κράτη για την περίοδο πριν το κράτασμό, πριν το σοκ, θα είναι επιλέξιμο σε αυτές οι χώρες να έχουν πρόσβαση. Έτσι θα αποφύγουμε το μυθικό κίνδυνο και θα δοθούν και περισσότερα κίνητρα συμμόρφωσης. Τι ενεργοποιεί τώρα την πρόσβαση. Αυτό θα πρέπει να είναι προκαθορισμένο. Παράδειγμα, τέτοια κριτήρια ενεργοποίηση θα μπορούσαν να είναι μεγάλες ε, και χρονοβόρες παρεκκλήσεις ε, των πολιτικών ή τάσεις ανεργίας ε, που επιμένουν το χρόνο. Αν λοιπόν πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας, θα είναι αυτόματη η παροχή υποστήριξης. Πρέπει να είναι αξιόπιστο και παρκές το μέγεθος αυτού του προϋπολογισμού. Άρα θα πρέπει να υπάρχει δανειοληπτική ικανότητα, ώστε να μπορεί να διαθέτει άμεσα πόρους αυτός ο μηχανισμός σταθεροποίησης. Θα καταθέσουμε προτάσεις πάνω σε αυτές τις γραμμές το Μάιο Τώρα είναι η ώρα να βράσουμε, έτσι πιστεύουμε. Οι διαπραγματεύσει θα είναι δύσκολε, αλλά νομίζουμε ότι υπάρχει περιθώριο ευκαιρία και είναι επίγον να, ολοκληρωθεί η Νομισματική Ένωση ω προ αυτό το σκέλο. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Σα ευχαριστώ. Πολύ πιστική συλλογιστική σας για τις ανάγκες που υπάρχουν για τη σταθεροποιητική λειτουργία αυτή. Το κρίσιμο είναι φυσικά πώς θα πετύχουμε αυτή τη λειτουργία. Περιμένουμε λοιπόν τις προτάσεις σας. Το μέγεθος όμως είναι ένα θέμα και φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν ερωτήσει. Και με ενδιαφέρει και αυτό που είπε ο κύριος Ρέγκλιν για το ESM, ότι μπορεί να είναι ένα ενδεχόμενο μηχανισμό διευκόλυνση, δεν ξέρω, να το πούμε μηχανισμό προστασία, backstop. <coughs> το σκέφτεστε αυτό ως ενδεχόμενο. Ή θα είναι τελείω διαφορετικά και ξεχωριστά ε, ως δύναμη πυρός αυτά τα δύο εργαλεία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τις παρεμβάσεις των μελών της Επιτροπής μας. Πρώτη ή πρώτος ο κύριος Όλμπριχτ. Α, έφυγε ο κύριος Όλμπριχτ. Και εκεί άτομα έφυγε. Κύριε Κέλμελ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ζητώ συγγνώμη, αλλά ήμουν μέχρι τώρα σε μια άλλη επιτροπή. Δεν παρακολούθησα λοιπόν το σύνολο της ομιλίας. Παρ' όλα αυτά ήθελα να ζητήσω το λόγο γιατί συνεχώς ασχολούμαι με το ζήτημα αυτό και πρέπει να ομολογήσω ότι όλα αυτά τα οποία ακούγεται είναι στον τομέα τη σφαίρα της θεωρίας και των συζητήσεων, αλλά η πράξη τα τελευταία χρόνια δείχνει εντελώ το αντίθετο. Και θα μπορούσε κανείς να αναφερθεί σε πάρα πολλές λεπτομέρειες, όπως παραδείγματος χάρη για το ESM, που δημιουργήθηκε ουσιαστικά ως κάτι προσωρινό, ως ένα μέτρο ε, δυσανάλογο και ασυνήθιστο κατά κάποιο τρόπο για την αντιμετώπιση μιας ανάλογης και ασυνήθιστης κατάστασης. Όταν λοιπόν ε, θα ήταν επιτυχής ο μηχανισμός αυτός μετά υποθέτει έπρεπε να καταργηθεί. Τώρα όμως βλέπουμε ότι ε, κατοχυρώνεται και γίνεται κάτι μόνιμο και αυτό πώς ε, ταιριάζει. Δεν ταιριάζει σε καμία περίπτωση. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη να, ότι κάτι δεν πήγε καλά. Ε, συνέχεια όμως ακούμε ότι είναι μια πολύ επιτυχημένη ιστορία το αλλά πρέπει να το σώσουμε συνεχώ από την άλλη πλευρά. Πάλι δεν ταιριάζουν αυτά μεταξύ του. Και πολλά είναι αυτά που δεν ταιριάζουν μεταξύ του. Κανόνε έχουμε. Υπάρχει η συνδίκη του Μαστρίχτ και εδώ και χρόνια σταμάτησαν να μετράνε όλοι πόσες φορές παραβιάζεται αυτή η συνθήκη. Γιατί δεν ενδιαφέρει κανέναν μάλλον το θέμα αυτό. Μπορούμε λοιπόν να, να ε, υιοθετούμε κανόνες και κανόνες. Έχουμε κανόνες που την πρώτη φορά που χρειάστηκε να εφαρμοστούν δεν ε, εφαρμόστηκαν. Επίσης κανόνες για τις τράπεζες. Ε, όταν τους ε, ορίσαμε, στην περίπτωση που έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά με τη Monte την Ιταλική τράπεζα, πάλι δεν τηρήθηκαν αυτοί οι κανόνες. Και τώρα λοιπόν συζητάμε πάλι για κανόνες πάρα πολύ αυστηρούς, αλλά κατά πόσον αυτό πρέπει να το πιστέψουμε, πραγματικά νομίζω ότι ξεκινάμε από λάθος αφετηρία δεδομένου του παρελθόντος. Και ούτε και η θεωρία ε, είναι σωστή. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα προστασίας, θα πρέπει ε, να υπάρχει και μία δέσμευση αυτό που θα συμμετέχει ότι θα συμπεριφέρεται με έναν σωστό τρόπο. Αν ξέρουμε όμως ότι σε πέτος ανάγκης ε, θα πληρώσει εν μέρει και κάποιο άλλο, μπορούμε να παίρνουμε πιο εύκολα κινδύνου. Ρίσκα μάλλον. Το ευρώ και τα κράτη ε, που συμμετέχουν θα πρέπει να, να φέρονται σωστά από δημοσιονομικής πλευράς. Ε, αλλά πραγματικά εγώ δεν καταλαβαίνω. Εδώ και πολλά χρόνια έχουμε τους κανόνες του Μαστρίχτα. Ε, αυτοί είναι οι κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται. Δεν χρειάζεται να υιοθετήσουμε νέους, αλλά να επιβάλλουμε την εφαρμογή των ήδη υφισταμένων. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριος Χέις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα σχολιάσω την εξαιρετική παρουσίαση του καθηγητού από την κλουκή περιφέρεια, αλλά πολύ ε, καλής παρατηρήσεις ε, του καθηγητού. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, μπορώ να κάνω εντελώς λάθος, αλλά ο πολιτικός που έχω μέσα μου μου λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμιά όρεξη για αλλαγή της συνθήκης και με βάση τις αναλύσεις που ακούσαμε για τη δημοσιονομική ικανότητα αναπόφευκτα θα πρέπει να υπάρξουν αυτές οι αλλαγές. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει πολιτική βούληση πρώτον και δεύτερον δεν είναι και σίγουρο ότι θα υπάρξει επαρκής υποστήριξη σε μια τέτοια ιδέα. Ο κύριος Νούνεθ ε, Φερέρ ε, είπε κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Είπε ότι η σταθερότητα ξεκινάμε πολύ καλά εθνικά συστήματα διαχείρισης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν εστιάσαμε παρκώς όμως ακόμη στην φυστάμενη αρχιτεκτονική στο πώς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, που δεν τα αντιλαμβάνονται όλα τα κράτη, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή δηλαδή των υφιστάμενων κανόνων. Δεν τα αντιλαμβάνονται τα κράτη μέλη όλα με τον ίδιο τρόπο. Αν δεν έχουμε λοιπόν ε, κοινού κανόνες που εφαρμόζονται, θα έχουμε προβλήματα. Μίλησατε και για το προπολογισμό. Εγώ τα θέτω αυτά τα θέματα συνεχώς. Πώς μιλήσατε για αυτή τη... το δόγμα, το 1% αν πρέπει να κλείσει η τρύπα του Brexit και αν θέλουμε να έχουμε συνεκτικό προπολογισμό μετά, αυτό το 1% το δόγμα ε, πρέπει να αλλάξει. Το δέχομαι και πρέπει να έχουμε ένα μεγαλύτερο προπολογισμό. Αλλά το σύστημα που έχουμε τώρα αυτό λέει, τι θα γίνει στο μέλλον δεν ξέρω. Σε αυτό το πλαίσιο όμως. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τον προπολογισμό για να πετύχουμε πολύ Περισσότερε και πιο συστηματικέ δημόσιε μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη. Και αυτό όχι μόνο ω κίνητρο για τον προπολογισμό, αλλά και για να υπάρχει αυτή η ισορροπία που είπατε εσεί ότι αφορά τη χρηστή διαχείριση. Δηλαδή θα πρέπει να είναι ένα κινητήρα, ένα μοχλός αυτό ο προπολογισμό για να υπάρχει συνεκτικότητα ε, και συνέπεια στι δημόσιε μεταρρυθμίσεις. Γιατί η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα είναι σίγουρα ένα ε, χρονοβόρο, μάλλον ένα δαπανηρό εγχείρημα, αλλά τον προπολογισμό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για πολύ μεγαλύτερες, βαθύτερες δημόσιες μεταρρυθμίσεις για να έχουμε αυτό που είπατε εσείς, δηλαδή βελτίωση της κατάστασης ε, σε επίπεδο κρατών μελών. Γκρέσλ Και εγώ έχω τις αμφιβολίες για το κατά πόσο όλα αυτά που ακούσαμε ταιριάζουν μεταξύ τους, για το, τα όσα ακούσαμε σήμερα. Για τον ηθικό κίνδυνο ρώτησε τον κύριο Ρέγκλινγκ. Στη Γερμανία μας απασχολεί πάρα πολύ το θέμα αυτό. Δηλαδή πληρώνουμε εμείς για αυτά που δεν θέλουν να κάνουν οι άλλοι. Και τελικά δεν έχουμε και καμία επιρροή στο τέλος. Πώς το βλέπετε εσείς. Ωραία τα λέμε εδώ και καθόμαστε Πώς τις βλέπετε εσείς ε, τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της ΕΚΤΑ και τι αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί με τώρα. Έχουμε ε, βελτίωση ή απλά τα έχουμε λίγο βάλει στην άκρη και μεταθέσει για μετά τα προβλήματα. Επίσης δεν έχω καταλάβει ακριβώς ε, πώς μπορούμε να τα παρουσιάσουμε όλα αυτά στους ψηφοφόρους μας. Φαντάζομαι θα βρούμε τον τρόπο αν είμαστε πεπισμένοι ότι είναι σωστό το πακέτο. Δεν είμαι ακόμα σίγουρη. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο προεπλογισμός της Ένωσης και πώς συνδέεται με τον προεπλογισμό για την Ευρωζώνη. Η Κομισιόν. Πώς βλέπετε τα μελλοντικά διαθωτικά ταμεία. Τι μέτρα θα προτείνει η Κομισιόν. ώστε τα κράτη τα οποία που παίρνουν αυτά τα χρήματα να τηρούν ε, αυτά που πρέπει να κάνουν. και δεν, είναι, δεν έχει συμπεριληφθεί ακόμη ο προπολογισμό αυτό στο συνολικό προπολογισμό τη Ένωση και αυτό με ανησυχεί. Και να ξέρετε ότι εδώ προβλέπεται συναπόφαση και υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να έχουν διαφορετικά σχέδια. Μπορεί ε, να υπάρξει πρόβλημα στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, Υπουργεία Οικονομικών, που έχουν συνηθίσει να θέτουν τα κονδύλια εκεί που θεωρούν ε, σκόπιμο. Δύσκολα ε, συντονίζονται όλα αυτά μεταξύ τους και δεν τα έχω καταλάβει πολύ καλά. Να μας τα διευκρινίσετε. Ευχαριστώ. Κύριος Μουρεσάν. εδώ στη γωνία. Τρεις ερωτήσεις στους τρεις ομιλητές. Καταρχάς, ποια είναι η σχέση ανάμεσα η νέα δημοσιονομική ικανότητα ή έναν προϋπολογισμό της Ευρωζώνης και τον σημερινό προϋπολογισμό της Ένωσης. Να το σχολιάσετε αυτό, γιατί στην Επιτροπή Προπολογισμών του Κοινοβουλίου μας απασχολεί η ενότητα του προπολογισμού. Ειδικά τα πρόσφατα χρόνια είδαμε πιστεύματα για την Αφρική, ε, το μηχανισμό διευκόλυνση για τους στην Τουρκία, το Μαντάτ, ε, είναι εκτό του προπολογισμού, εκτό του πλαισίου αυτού της Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερη ερώτηση είναι το μέγεθο αυτή τη δημοσιονομική ικανότητα και πώ θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί. Υπήρξαν κάποια σχόλια που ακούσαμε και μα έδωσαν κάποιες ιδέες ε, τι παρουσιάσει που ακούσαμε, αλλά θα θέλαμε λιγάκι περισσότερες διευκρινήσει. Πόσα λεφτά θεωρείτε ότι χρειάζονται για αυτή τη δημοσιονομική ικανότητα και ποιε είναι οι πηγέ χρηματοδότηση. Τρίτον, Ποιο είναι ο ρόλος για το Κοινοβούλιο, ε, για τη διακυβέρνηση ενό τέτοιου μηχανισμού δημοσιονομική ικανότητα ή ενό προπολογισμού τη Ευρωζώνη. Ευχαριστώ. Thank you. Um, Ευχαριστώ. Α υποφεληθώ κι εγώ. Α, βεβαίω και εσεί και εσεί, κυρία Μπερέ. Uh, ε, okay, to... η κυρία Μπερέ, θα προσπαθήσω να μιλήσω γαλλικά. Όχι, σα παρακαλώ. Εγώ προεδρεύω, σα δίνω το λόγο όταν θέλω. Θα τον πάρετε το λόγο, αλλά όχι τώρα. Υπάρχει και κατάλογος. Κυρία Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Νουνές που αναφέρατε τους ισολογισμούς και την δυνατότητα διαχείρισης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Έχουμε συνεχώς προβλήματα με την αξιολόγηση των μη οικονομικών στοιχείων του προπολογισμού. Ε, θα πρέπει να διαχειριζόμαστε τα στοιχεία ακόμη και όταν δεν είναι οικονομικής φύσεως, στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, έτσι. Θα πρέπει να δούμε τι είναι η καθαρή αξία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο επιμέρου κρατών μελών πάνε πάνω, πάνε κάτω, γιατί αυτό δείχνει κατά πόσο υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη ή όχι. Το μήνυμά σα όμω είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί με το μικρό προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω είπατε, δεν μπορούμε να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα. Χρειαζόμαστε συνέργειε με του εθνικού προπολογισμού. Πώ θα δημιουργήσουμε αυτέ τι συνέργειε με του εθνικού προπολογισμού, ειδικά όταν μιλάμε για μια δημοσιονομική ικανότητα. Και να ρωτήσω και εγώ κάτι που ρώτησαν και οι άλλοι συναδελφοί. Το 1%, το ανώτατο όριο του 1% είναι η οροφή. Ε, όμως η Κομισιόν έχει αυτή την πρόταση 1,1 χ. Και εμείς έχουμε κάνει την πρόταση 1,3. Έτσι. Για, για τον προβλησμό της Ένωσης. Αρκεί όμως για να αποκτήσουμε αυτή τη δημοσιονομική ικανότητα που χρειαζόμαστε. Ε, Επίσης υπόθηκε από τον ομιλητή ότι αυτή η δημοσιονομική ικανότητα θα πρέπει να εστιάζει περισσότερο στην Ευρωζώνη. Δεν μπορούμε να έχουμε ισχυρή, ισχυρή Ευρωζώνη χωρίς ισχυρά κράτη-μέλη εκτός της Ευρωζώνης που συγκλίνουν προς την Ευρωζώνη γιατί είναι τμήμα της εσωτερικής αγοράς και αν δεν είναι δυνατά και αν δεν, δεν υπάρχει ε, καλή αγορά η οποία θα εισάγει από την Ευρωζώνη, ας πούμε, πώς θα δημιουργήσει ένα ωραίο και συνεκτικό όλο όλα αυτά. Και για τον κύριο Φαμπρίνη αναφέρατε ότι θα πρέπει να αποφύγουμε τις μεταφορές πιστώσεων από κράτος σε κράτος. Τι, οποιοδήποτε είδους ε, μεταφορές, ναι μεν, αλλά υπό ώρες. Σας παρακαλώ να το σχολιάσετε λίγο παραπάνω για να το καταλάβω. Thank you. Ευχαριστώ. Και τώρα κυρία Uh, ε, θα μιλήσω γαλλικά. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον. Σα ευχαριστώ για τι συνεισφορέ σα, για τι ομιλίε σα και τι παρουσιάσει σα Να θέσω δύο-τρία ερωτήματα. Ο Κλάους Ρέγκλινγκ μας είπε ότι οι σημερινοί κανόνε επιτρέπουν να ανταποκριθούμε σε συμμετρικά σοκ. Αυτό είδαμε την περίοδο 2009-2010. Και ένας άλλος ομιλητής, η Ανιές, είπε ότι είχαμε επαρκείς κανόνες, η Ανιές Βενέση και ότι δεν χρειαζόμαστε ένα πολύ μεγάλο συμπληρωματικό προϋπολογισμό. Εντάξει. Εγώ όμως δεν συμμερίζομαι αυτή την ανάγνωση της ιστορίας. Έχω την αίσθηση ότι η απουσία επαρκούς περιθωρίου το 2009 και 2010 για να αντιμετωπίσουμε τα συμμετρικά σοκ λόγω κρίσης οδήγησαν σε αυτό που υπενθύμησε η Κομισιόν που ήταν ε, μία κρίση ή μία ύφεση αυτοτροφοδοτούμενη που φτιάξαμε εμείς οι ίδιοι την περίοδο 2012 με 2015. Άρα θα πρέπει να ξαναδούμε τους κανόνες. Επίσης, η ιδέα. Μία ερώτηση προς τον κ. Νιουνιές Φερέρ. Δεν συμφ συμμερίζομαι με όλες τις ιδέες σας. Είπατε όμως ότι αυτό που δεν κοιτάμε είναι πώς διαχειρίζονται τον προπολογισμό του στα κράτη-μέλη. Συμφωνώ. Το καταλάβαμε και με την Ελλάδα όταν στείλαμε μία ομάδα εργασίας αυτή την περίφημη task force για να εξηγήσουν στους Έλληνες πώς πρέπει να διαχειρίζονται τον προπολογισμό τους και τα δημόσια οικονομικά τους. Αλλά πρέπει να διδαχθούμε από αυτήν την ιστορία. Αυτό σημαίνει ότι οι κανόνε τη διακυβέρνηση και του συμφώνου σταθερότητα δεν, είναι δεν είναι καλοί. Δεν ε, έχουμε του καλού δείχτε. Ή δεν βάζουμε τον νι, ας πούμε, στα καλά τετραγωνίδια, ας πούμε, ε, σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά των κρατών μελών και πρέπει να είμαστε σοβαροί. Και πρέπει να ξέρουμε ότι ο προπολογισμό τη Ένωση θα πρέπει να υποστηρίζει το διοικητικό δυναμικό των κρατών μελών αλλά το διοικητικό δυναμικό που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη με κλασικό τρόπο θεωρείται στο Συμβούλιο ότι έχει φοβερούς κινδύνους διαφθοράς. Πώς επιλύουμε την αντίφαση αυτή. Κλάους Ρέγκλινγκ. Άλλη μια ερώτηση, μετά από αυτά που είπε και η Κομισιόν για την ε, λειτουργία της σταθεροποίησης. Δεν ξέρω αν αυτά που παρουσιάστηκαν θα είναι το τελικό αποτέλεσμα στις 29 Μαΐου. Εάν ναι, είναι καλή, καλός ιονός. Δεν θέλω όμως ε, να ξεχνάμε ότι έχουμε όλα τα κριτήρια, να περάσουμε τους επιτρόπους και τα λοιπά, να περάσουμε τους προέδρους των επιτροπών. Αν περάσει όμως, τότε υπάρχει μία σχέση ε, για να, με το ESM, με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, μία δυναμική σχέση. Πώς βλέπετε, ας πούμε, την εξέλιξη του δικού σας οργάνου μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και άλλα δύο σχόλια, αφού σας άκουσα όλους. Αν είμαστε σε ένα ιδεατό κόσμο, οι περισσότεροι ομιλητές θα ορκιζόντουσαν ότι ο καλύτερος τρόπος σταθεροποίησης είναι η... ένα ελάχιστο επίδομα ανεργίας. Το λέει το Δουνουτού επί χρόνια. Ο Ρέιμαρ Μπέργκη και εγώ δεν συμφωνήσαμε τελικά για το θέμα αυτό, ελάχιστο επίδομα ανεργία. Αν ξεπεράσουμε όμω το θέμα των εμποδίων κτλ., αν ρωτήσουμε του εμπειρογνώμονε, το ένα τέλειο ε, πλαίσιο σταθεροποίηση δεν θα ήταν ένα ελάχιστο επίδομα ανεργία. Τέλο, να υπενθυμίσω ότι το να μετασχηματιστεί ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο για να γίνει κάτι τέτοια ε, θα πρέπει να δοθεί μια μάχη. Θα πρέπει να την κερδίσουν αυτοί που είναι υπέρμαχοι τη μετατροπή. Εμένα με ενοχλεί λιγάκι, αλλά τέλο πάντων ε, έκανα μια υποχώρηση απέναντι στον κύριο Μπέγκε και δεν θέλω να την πάρω πίσω. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να τη γράψουμε το δούνου του και να, να κάνουμε ένα αντίστοιχο πράγμα για το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Γιατί υπάρχουν καταρχά ο βαθμό ολοκλήρωση, το δημοκρατικό πλαίσιο εκπώνηση των οικονομικών πολιτικών δεν, δεν είναι ίδιε ανάμεσα στο Δουνουτού και το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Άλλο η Ευρωζώνη, άλλο οι χώρε που παρεμβαίνει το Δουνουτού. Έπειτα, οι διατάξει του άρθρου 4 του Δουνουτού για την κατάσταση των κρατών δεν μπορεί να μεταφερθεί στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, γιατί τότε θα. Αντι... Ε, θα... Αυτό δεν θα ήταν σύμφωνο με τι συνθήκε. Και τελευταίο σημείο που δεν υπάρχει στο Δουνουτού είναι ότι έχουμε ένα ευρώ και έχουμε ε, τη δυνατότητα ε, σοβαρής εποπτείας των αγορών. Τη δουλειά που κάνει το SSM και το SRB. Αυτά ελπίζω να κάλυψω όλα τα στοιχεία. Και τώρα ο κ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω κι εγώ. Έκανα κάποιες ε, υποχωρήσεις, ε, αλλά μετά από τη σημερινή συζήτηση η έκθεση αυτή νομίζω έθεσε τα θέματα τα πολύ σημαντικά ίσως νωρίτερα από άλλες επιτροπές ε, ή από άλλα φόρα. Πριν από 14 ημέρες είχα μια εκδήλωση με το εμπορικό και μηχανικό επιμελητήρια στη γερμανική μεθόριο και από ένα κολέγιο από το Αμβούργο, από το Europa College, είχαμε ένα συνάδελφο ε, που μας ε, μίλησε λόγω και το ότι είμαστε στα σύνορα με τη Δανία ότι δεν χρειαζόταν η Δανία. Δεν χρειαζόταν κοινό νόμισμα ουσιαστικά λόγω ε, της ε, κοινή αγοράς. Είμαι 51 ε, και έχω ζήσει πολλά και πολλά και τις αναταραχές ε, που ζήσαμε τότε στα κράτη-μέλη με τις συνεχείς υποτιμήσεις των νομισμάτων ε, με, τεράστιες, ε, με τεράστια προβλήματα και αυτό ήταν η βάση για όλα τα βήματα τα οποία έκτοτε ακολούθησαν. Αν μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση, γι' αυτό έκανα λόγο πριν για προβλεπτική, για proactive πολιτική, παραδείγματος χάρη, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη μεταναστευτική ε, πρόκληση και Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που έχουν στυλώσει τα πόδια τους και όταν είχε προκύψει η μεταναστευτική κρίση δεν ήθελαν να δημιουργηθεί αυτός ο μηχανισμός για παραδείγματο χάρη την κοινή συνοριοφυλακή. Και έλεγαν αρνούμαστε, δεν το θέλουμε αυτό όπως η Γάλλη για παράδειγμα. Όταν όμως υπήρξαν απρόβλεπτες εξελίξεις στον κόσμο, γιατί στον κόσμο υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι και δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε όλα και τη βλέπουμε ότι πιανόμαστε απροετοίμαστοι. Υπάρχει ε, στην σύμβαση μια πιστοτική διευκόλυνση, αλλά για κράτη, κράτη που δεν είναι μέλη ε, της Ένωσης. Λες και θεωρούσαμε ότι στην Ένωση θα είναι όλα τέλεια. Άρα θα πρέπει ε, τώρα να καταλάβουμε ότι πρέπει να λάβουμε και προληπτικά μέτρα και να δείξουμε και προς τα έξω ότι είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε τις αξίες, της αρχές μας, την εσωτερική αγορά, το κοινό νόμισμα, το ευρώ. Αυτά πρέπει να τα υπερασπιστούμε, να τα προσπατεύσουμε με οποιοδήποτε ε, συνέπεια αυτό συνεπάγεται. Και σε σχέση με αυτά τα οποία είπε η Περβάνσε, σε σχέση ε, με τον κύριο Ρέγκλη και την κυρία Μπενασί, ε, για την ε, δημοσιονομική δυνατότητα έχουμε αναφέρει πώς θα χρηματοδοτηθεί διάφορες εναλλακτικές, διάφορα σενάρια Μπορεί να γίνει με εισφορές από τα κράτη-μέλη, χρηματοδότηση μπορεί να γίνει με, τις, ε, με τα έσοδα, ε, above the ceiling of the ESM και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα εθνικά κοινοβούλια επίσης ε, θα πρέπει και αυτά να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε σε όλα τα επίπεδα τον κοινοβουλευτισμό, άρα θα πρέπει να υπάρχει έλεγχο, και πρέπει αυτός ο έλεγχο να δοθεί στα χέρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν γίνει λόγο και για το ασφαλιστικό μοντέλο. Πριν από ένα χρόνο λοιπόν στην έκθεσή μας είχαμε εκφράσει αυτή την ε, <clears throat> προϋπόθεση, χωρίς να έχουμε βέβαια συμφωνήσει, αλλά είχαμε πει ότι θα πρέπει να υπάρξουν σημαντικές ε, βελτιώσεις και μιλήσαμε για το μέγεθος ε, και για τον τρόπο χρηματοδότησης και είπαμε ότι θα πρέπει να είναι ουδέτερο δημοσιονομικά για ένα μακροχρονικό διάστημα. Αυτό ήταν ε, η συμβιβαστική πρόταση στην οποία μπορέσαμε να καταλήξουμε επειδή θέλουμε να είναι σταθερή κατάσταση. Τώρα, πάντα για τον κύριο Ρέκλινγκ μίλησε για ένα βράχυπρόθεσμο δανεισμό από το ESM με πιο ελαφρύς όρους. Από πλευράς οικονομικών υπάρχουν κάποια ζητήματα, ασφαλιστικό μοντέλο, εισφορές και η δυνατότητα να χρησιμοποιούμε το ESM ή το νομισματικό ταμείο. Η αιρεσιμότητα ήταν ένα θέμα που συζητήσαμε, οι αιρεσιμότητε μάλλον. Και έχουμε και τις συζητάσεις αναχώρα. Θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε και στο πλαίσιο το συζήτησης για τα ταμεία συνοχή και τα διαρθρωτικά ταμεία. Παίζουν ένα ρόλο. Το θέμα είναι η βιώσιμη σταθερότητα. Και αυτό σε σχέση με αυτά που και ο κύριος Νιούνιες φέρεται, έχει να κάνει με τη δημοσιονομική διαχείριση των ε, κρατών μελών. Αν απαιτήσουμε όμως ακριβώς αυτό, νομίζω από τα κράτη-μέλη μου δημιουργείται το ερώτημα μήπως αυτό που λέγαμε εμείς ε, για τις προϋποθέσεις ε, και τις τους όρους ή έναν λεγόμενο κώδικα σύγκλησης. Μήπως αυτό θα ήταν κάτι που σχετικά θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Αυτά, ευχαριστώ. Thank you. Jean ευχαριστώ, Jean Ευχαριστώ, Ρομπέρτο. Να πω πρώτα απ' όλα ότι Δυστυχώς δεν ήμουν εδώ την πρώτη ώρα ε, και λυπάμαι γι' αυτό. Είχα μια άλλη δεσμασή και δεν μπορούσα να τη μετακινήσω. Ευχαριστώ και τον κύριο Μουρεσάν που με αναπλήρωσε. Ε, έχουμε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα μπροστά μας, την διακυβέρνηση της Ευρωζώνης. Έχουμε περάσει στο ενιαίο νόμισμα λόγω των ανταγωνιστικών υποτιμήσεων που διακύβευαν την ενιαία αγορά και έχουμε επηρεάσει την ε, ανάπτυξη, μπορεί να αυξηθεί και η ανεργία στην Ευρώπη. Αλλά εάν κατορθώσαμε να έχουμε μια ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική ε, Τράπεζα, αφήσαμε τη διακυβέρνηση στα χέρια των κρατών μελών. Από τη μια πλευρά έχουμε μια ενιαία νομισματική πολιτική, αλλά έχουμε ε, εθνικές οικονομικές πολιτικές συσσωρευμένες και δεν έχουμε τη, δυνατότητα να κάνουμε αυτό το policy mix που γίνεται στη ΣΥΠΑ, για παράδειγμα. Και δεν βλέπω πώς θα μπορέσουμε να επιλύσουμε το θέμα αυτό με την, τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα της Ευρωζώνης, γιατί όταν δημιουργήθηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, όταν έπρεπε να δοθεί το κεφάλαιο, δεν ήταν τα 28 κράτη-μέλη που συμμετείχαν, ήταν τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Όταν χρειάστηκε να δοθούν εγγυήσεις για να ε, δοθούν δισεκατομμύρια στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό ε, Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δεν ήταν τα 28 μέλη που δώσαν την εγγύηση, αλλά τα μέλη της Ευρωζώνης. Άρα αυτό δημιουργεί μια ευθύνη, ιδιαίτερη ευθύνη, που θα πρέπει να μας οθήσει, ε, να μας δώσει περισσότερη ε, ισχύ στην ε, διαχείριση. Είχαμε την ευκαιρία να, είχαμε μια, να δημιουργήσουμε μια αποστολή βοήθειας για την Ελλάδα και όταν οι Έλληνες συνάδελφοι όταν βλέπουν την πραγματικότητα των, αριθμών, το, το γεγονός ότι δεν είχαμε πιο ισχυρή αντίδραση αν έχουμε μια κοινή μοίρα. Α συμφωνήσουμε πώς θέλουμε να παρουσιάζουμε τους δημόσιους υπολογισμούς; τους ε, ε, άρα μερικές φορές θα πρέπει να έχουμε λίγο, λίγο πιο έντονες σχέσεις και να πούμε αρκετά ε, σταματήστε να ακολουθείτε τον κύριο Γεωργίου που τελικά πήγε στη Washington για να γλιτώσει από τις κυρώσει ε, της ελληνικής δικαιοδοσίας. Αυτού του λεχθέντος τώρα. Ε, ποιος είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Ε, οι συνθήκες δεν μας επιτρέπουν να ακολουθήσουμε κάποιες κατευθύνσεις, αλλά έπρεπε να πούμε τι πρέπει να θεσπίσουμε, να φτιάξουμε και να δούμε και τη δημόσια γνώμη, να ασκήσουμε πίεση στους αρχηγούς κρατών, έτσι ώστε να αλλάξουν οι συνθήκες. Έπρεπε να δούμε τι ε, θα έπρεπε να ήταν η διακυβέρνηση της Ευρωζώνης. Τελευταία ερώτηση προς τον Κλάουσερ Έγκλινγκ. Ε, μόλις τώρα διάβασα το κείμενό του, την παρουσίασή του και βλέπω μια παρατήρηση πολύ ενδιαφέρουσα γιατί ε, λέει ότι ε, πρέπει να μελετήσουμε τα public goods, τα λεγόμενα δημόσια αγαθά δηλαδή την προστασία των συνόρων, την, των εξωτερικών συνόρων, ένα σύστημα κοινή άμυνας, μέτρα κατά της αλλαγής του κλίματος, εάν ενσωματώσουμε αυτά τα δημόσια αγαθά στον ευρωπαϊκό προπολογισμό, κύριε Ρέγκλινγκ. Δεν πρέπει να φανταστούμε αν το κάνουμε αυτό είναι γιατί τα κράτη-μέλη ε, δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικά σε ε, εθνικό επίπεδο για αυτά τα δημόσια αγαθά και δεν ήρθε η ώρα να καλέσουμε τα ε, κράτη-μέλη να ενσωματώσουν αυτά, αυτές τις δαπάνες στον προπολογισμό έτσι ώστε να έχουμε έναν ευρωπαϊκό προπολογισμό που να αυξάνεται χωρίς να αυξάνονται και οι δαπάνες. Thank you. Σας ευχαριστώ. Έχω και εγώ μια-δύο ερωτήσεις προς τους ομιλητές μας. Βάσει της ε, κοινή ε, συμφωνίας συνένεσης έχουμε πολλά εργαλεία, πράγματι. Αυτό που μας λείπει είναι η μακροοικονομική σταθεροποίηση απέναντι στα ασύμετρα σοκ. Και βλέπω ότι υπάρχει συμφωνία, ιδιαίτερα σε αυτά που ανέφερε ο κύριος Ρέκλη και η Κομισιόν. Καταρχάς, όπως είπε και η Μπερμπάνς, θα ε, να δω αυτά που είπε ο κύριος Ρέγκλινγκ. Έχουμε χώρο, περιθώριο ελιγμού ε, κατά των ε, ασυμμετρών σοκ. Το είδαμε το 9 και το 10. Το, είναι σημαντικό ότι το τι έγινε το 11, το 2011 δημιουργήσαμε περισσότερα σοκ παρά ε, αυτά που απορροφήσαμε λόγω πρώτα απ' όλα της έλλειψης προληπτικών εργαλείων και κατά δεύτερο λόγο ενός συνδυασμού του συνδρόμου Ντοβίλ, της δημιουργίας ε, αυτών των κινδύνων. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε αυτόν τον συνδυασμό της Ντοβίλ και της ε, προκυκλικής ε, δημοσιονομικής εξυγίανσης. Αυτό πυροδότησε μια δεύτερη κρίση και γι' αυτό ξεπεράσαμε το ΕΠΑ από αυτό του, τον είπα γιατί, γιατί έχουμε μια δεύτερη κρίση και τα εργαλεία μας δεν ήταν ικανά να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση. Είχαμε πρώτα απ' όλα την ε, Ντοβίλ και την δημοσιονομική ε, εξυγίανση και για να διορθώσουμε αυτήν την κατάσταση δημιουργήθηκαν προβλήματα διότι είχαν ασκήσει υπερβολικές πιέσεις στην δημοσιονομική πολιτική και την οικονομική πολιτική, νομισματική πολιτική. Εάν είχαμε προληπτικό μακροοικονομικό εργαλείο σταθεροποίησης θα μπορούσαμε να αποφύγουμε και την καταστροφή της Ντοβίλ και την λιτότητα αλλά και την ε, άσκηση πίεσης στις, στους δημοσιονομικούς κανόνες και την νομισματική πολιτική. Εάν αυτό αληθεύει, αν υπάρχει ε, συμφωνία σε αυτή την ανάλυση, υπάρχουν δύο θέματα. Θα ήθελα να ρωτήσω κυρίως τον κύριο Ρέγκλινγκ και τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Πρώτον, Εάν θέλουμε να αποφύγουμε την επίδραση Ντοβίλ, είναι απαραίτητο να πάρουμε οτιδήποτε ε, μπορεί να προκαλεί στο στρες στην αγορά, ακόμη και αν γίνεται για να δημιουργηθεί μια καλύτερη πειθαρχία των αγορών που θα μας βελτιώσει. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν βλέπω ότι είναι πιστική η έκθεση, γιατί φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει αντάλλαγμα ανάμεσα σε περισσότερο λιγμό σε εθνικό επίπεδο. Νομίζω θα πρέπει να κάνουμε το αντίθετο. Να δούμε μεγαλύτερη σύγκληση και αιρεσιμότητα προς σύγκληση. Εάν αυτό ισχύει και η Κομισιόν δεν έχει θέσει μηχανισμούς αναδιάρθρωσης. Τι, έχει, τι εννοείτε όταν λέτε ότι πρέπει αυτές οι διαπραγματεύσεις να γίνουν πιο συστηματικές και προβλέψιμες, διότι όπως είπατε εσείς σωστά, ήδη έχουμε τη δυνατότητα ε, για την αναδιάρθρωση των δημοσίων ε, δανείων. Ε, θα ήταν λάθος να, κάνουμε, να το κάνουμε ως υποχρέωση. Είναι κάτι το οποίο δεν θα λειτουργήσει ποτέ. Ε, το αποκλείουν τα κράτη-μέλη. Δεν είναι θέμα αυτό που τίθεται επιτάπητος. Αλλά πραγματικά θα βοηθούσε να έχουμε μια πιο συστηματική διαδικασία όταν χρειάζεται να γίνει αναδιάρθρωση. Πώς βλέπετε όμως τη διαφορά ανάμεσα στο προβλέψιμο και το αυτό ε, υλοποιήσιμο. Θα μπορούσατε να το αναπτύξετε αυτό το θέμα. Το δεύτερο, αυτό που είπατε κύριε Ρέκλινγκ, για τη δυνατότητα το ESM να έχει μια, ένα νέο μέσο δημοσιονομικό για τη μακροοικονομική σταθερότητα. Αυτό είναι ε, πολλά υποσχόμενο. Αν δεν αυξήσουμε σημαντικά τον προπολογισμό, ε, δεν ξέρω πώς θα μπορεί να επιτελεστεί αυτή η λειτουργία μέσα στα όρια του τρέχοντος προϋπολογισμού. Δεν ξέρω πού θα βρούμε το δημοσιονομικό χώρο ε, με αυτό το προπολογισμό, το τρέχοντα. Υπάρχει κάποιο χάσμα ανάμεσα στην ανάλυση της Κομισιόν και αυτό αυτό που θα συμβεί. Άρα, μπορούμε να φανταστούμε μια τέτοια λειτουργία μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού για τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη, όπως είπε και ο κύριος Μπέγκε, που να αποτελεί ένα δίκτυο χρηματοπιστωτικής ασφάλειας αλλά αυτό δεν θα απαιτούσε να ενσωματώσουμε το ESM μέσα στο νομικό πλαίσιο. Γιατί τα κράτη-μέλη αποφασίζουν πρώτα να δουν το περιεχόμενο και μετά να δουν εάν πώς θα προχωρήσουμε. Δεν ξέρω αν είναι πολύ καλή ιδέα αυτή. Δεν το 352 δεν ξέρουμε ακόμη αν υπάρχει, είναι μια πρόταση της Κομισιόν. και δεν ξέρω αν η Κομισιόν ήδη παρέχει στήριξη σε διακυβερνητικό επίπεδο. Άρα πρέπει να αποφασιστεί επιτέλους αυτό και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να μην μας αποτρέπει στο να κάνουμε αυτό τον δυνητικό συνδυασμό για να ε, κάνουμε ε, πιο βιώσιμη την δημιουργία αυτής της ε, λειτουργίας. To reconcile the other things we need to do, the borders, the defense, the the, the, of funds, the agriculture, the uh, Έχουμε όλα τα ταμεία, τα διαρθρωτικά κλπ. και Ακόμη και αυτό το 1,3% θα είναι πρόκληση. Αλλά δεν ξέρω αν δεν ε, ενσωματωθεί το ESM μέσα στο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν βλέπω πώς αλλιώς μπορεί να επιληφθεί. Αυτές είναι ερωτήσεις προς τους ομιλίες. Κύριε Ρέγκλινγκ, θέλετε να απαντήσετε. Ναι. μου δίνετε μια ώρα να απαντήσω τώρα. Να προσπαθήσω όσο πιο γρήγορα να απαντήσω. Πολλές διαφορετικές ερωτήσεις. Κυρία Γκρέσλερ, ρωτήσατε για τον ηθικό κίνδυνο. Δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα ε, με τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Η αιρεσιμότητα υπάρχει για να αποτρέψει το moral hazard και είναι τόσο αυστηρή αυτή η αιρεσιμότητα, αυτή, αυτές οι προποθέσεις τόσο αυστηρές, λένε ορισμένοι, που καμία κυβέρνηση δεν πρόκειται να ζητήσει δάνειο κατά πάσα πιθανότητα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Ε, θα υπάρχει επίσης και κάποια κριτήρια επιλεξιμότητας ή ρεσιμότητας ε, για να υπάρξει στήριξη στα πλαίσια της δημοσιονομικής σταθερότητας, για τη δημοσιονομική σταθερότητα. Πολλοί από εσά ρωτήσατε τα θέματα της, τα της δημοσιονομικής ε, σταθερότητας. Ο κ. Μόρισον ρώτησε τη σχέση που έχει ο προπολογισμός της Ένωσης και με αυτή την δημοσιονομική ικανότητα, ποιο είναι το μέγεθος, ποια η πηγή της χρηματοδότησης. Φυσικά το θέμα είναι πώς οργανώνεται. Υπάρχουν διαφορετικά εργαλεία για να πετύχουμε την μακροοικονομική σταθεροποίηση. Πολύ αναφέρατε, ας πούμε αυτό το Ταμείο για τις δύσκολες μέρες, ε, ένα συμπληρωματικό μηχανισμό ε, επιδόμου ανεργία, όχι πλήρη εναρμόνιση, συμπληρωματικό μηχανισμό τύπου ΙΠΑ, όπου υπάρχει μια πιστοτική γραμμή για τις πολιτείε που έχουν ειδικά προβλήματα, ω οικονομολόγο μου φαίνεται ενδιαφέρον. Καταγράφω ότι στην πολιτική συζήτηση όμως ε, αυτό το θέμα όλοι το βλέπουν αρνητικά. Γι' αυτό βλέπουμε να ψάχνουμε όλοι διαφορετικές ε, βραχυπρόθεσμες, ας πούμε, εναλλακτικέ. Ε, να δίνουμε δάνειο όχι για 20-30 χρόνια, αλλά για 4-5-6 χρόνια και να πληρώνονται μέσα στα πλαίσια του ίδιου οικονομικού κύκλου. Αυτό πολιτικά μπορεί να είναι πιο αποδεκτό. Θα μπορούσα όμως να συζητήσω και ένα σύστημα επιδομάτων ενεργείας. Ίσως πολιτικά και οικονομικά είναι ευκολότερο. Γιατί υπάρχουν οι προϋποθέσεις, πολλές από τις προϋποθέσεις ήδη. Ένα άλλο σημαντικό θέμα, όταν κοιτάξετε τον προπολογισμό της Ένωσης σε αντιδιαστολή με τη δημοσιονομική ικανότητα, κατά την άποψή μου, πού είναι το χάσμα και προσπάθησα να το εξηγήσω, είναι ότι χρειαζόμαστε αυτή την μακροοικονομική δυνατότητα σταθεροποίησης για να απορροφά τα σύμμετρα σοκ. Ε, κάτι διαφορετικό από τον προπολογισμό της Ένωσης, είναι, μιλάμε, μιλάμε για ένα κουμπαρά, ας πούμε, ένα εκπεριτροπής ταμείο που κάποια χρόνια κανένας δεν το χρειαστεί, αλλά όταν υπάρχει ένα σοκ, ας πούμε, ή διαφορές στις οικονομίες των διαφόρων κρατών της Ένωσης, της Ευρωζώνης μάλιστα, θα χρειαστεί αυτός ο κουμπαράς. Γι' αυτό δεν είναι αιτήσιος προπολογισμό. Και αυτό το διαφοροποιεί πάρα πολύ ε, όταν πάμε στη συζήτηση της χρηματοδότησης. Ε, είναι τελείω διαφορετικό από την περίπτωση του ετήσιου προπολογισμού και του πώ χρηματοδοτείται αυτό. Απάντησα στι ερωτήσει Μπέγκε για το πλαίσιο. Ε, συμμετρικά σοκ. Πολλοί από εσά αναφερθήκατε σε αυτό που είπα εγώ, ότι δεν θεωρώ ότι υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία ε, ενός δυναμικού που θα αντιμετωπίζει τα ασύμετρα σοκ. Το θέμα είναι πώς ερμηνεύουμε τις εξελίξεις ανάμεσα στο 2008 και 2015, ας πούμε χοντρικά σε αυτήν την περίοδο. Αρχικά δεν υπήρχαν προκυκλικές πολιτικές. Ε, η Αγνιές είπε ότι πάντα βλέπουμε προκυκλικές δημοσιονομικές πολιτικές, αλλά εγώ δεν το θεωρώ σωστό αυτό. Ε, η απάντηση στην παγκόσμια οικονομική κρίση οδήγησε σε αντικυκλικές πολιτικές ε, σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό πλαίσιο. και από 0,5% ε, έφτασε στο 6% το δημοσιονομικό έλλειμμα, ας πούμε. Και το, ε, το χρέος της Ευρωζώνης έφτασε, ε, ανέβηκε κατά 35% ας πούμε του ΑΕΠ. Αν είχαμε τέτοιες πολιτικές, αν είχαμε προκυκλικές πολιτικές, νομίζω ότι θα είχαμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Προσοχή λοιπόν στις ερμηνείες. Επίσης, ε, διάφωνησα με κάποιον με τον οποίο συμφωνώ συνήθως. Α, όταν συγκριθούμε με τη ΣΥΠΑ, ε, και λέτε ότι είπα ήδη το 2011 ε, φτάσανε στα επίπεδα του ΑΕΠ που είχαν πριν την κρίση, ενώ εμείς στην Ευρωζώνη τέσσερα χρόνια αργότερα, διαφωνώ. Μην ξεχνάτε ότι η ανανέωση πληθυσμού στην, στη ΣΥΠΑ ε, είναι πολύ ψηλότερη από την Ευρώπη. Μισό τα εκατό το χρόνο. Και θα πρέπει να κάνει τον υπολογισμό ε, του κατακεφαλήν ΑΕΠΑ για να δούμε πώς ε, εξελίσσεται το βιωτικό επίπεδο. Και οι συγκρίσεις είναι πολύ διαφορετικές, γιατί οι ΙΠΑ ε, αναπτύσσονται μισό τα εκατό γρηγορότερα το χρόνο για να έχουν ε, το ίδιο επίπεδο βιωτικό που έχουμε στην Ευρώπη. Προσοχή, προσοχή με τη σύγκριση. Η Ευρώπη δεν τα πάει και τόσο χάλια ε, με τις δύο κρίσεις που είχαμε. και αυτή είναι η διαφορά με τη ΣΥΠΑ, γιατί είχαν μόνο μία κρίση, όμως είχαμε δύο. Ε, από το 2016 όμως, 2016-2017, αλλά και το φέτος και του χρόνου, ε, θα έχουμε υψηλότερη αύξηση του ΑΕΠ από τη ΣΥΠΑ. Τέσσερα χρόνια θα έχουμε υψηλότερη ανάπτυξη του ΑΕΠ από τη ΣΥΠΑ. Ε, το χρειαζόμαστε γιατί πρέπει να πιάσουμε τη ΣΥΠΑ. Και τώρα πάω στον κύριο Αχτουή και σε ερωτήσεις του. Συμφωνώ μαζί σας εάν τα καθήκοντα φύγουν από τον εθνικό προπολογισμό και πάνε στον ενωσιακό, θα πρέπει να υπάρξει και κατάλληλη χρηματοδότηση. Συνολικά δεν θα πρέπει να αλλάξει η κατάσταση των ελλημάτων. Ο Ρομπέρτο Γουατιέρη. Κοίταξε τι κάναμε στις δύο κρίσεις που περάσαμε, έκανε έναν απολογισμό. Νομίζω είναι δύσκολο να ξεμπλέξουμε τις δημοσιονομικές επιπτώσεις και αυτό που προκαλέσαμε οι ίδιοι, ας πούμε, όταν μίλησα για την ανάγκη να γίνει η αναδιάρθρωση του χρέους πιο προκλέψιμη και πιο διαφανής, ο σκοπός είναι για να αποφύγουμε ε, δεύτερη διπλή ύφεση, ας πούμε. Δεν μιλάω για ένα μηχανισμό λοιπόν, γι' αυτό μιλάω για πλαίσιο, χωρίς αυτόματους κανόνες, καμία, κανένα αυτοματισμό στην, στην αναδιάρθρωση. Θέλουμε να ξέρουμε όμως, τι όλοι να ξέρουμε τι θα συμβεί αν συμβούν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό δεν συμβαίνει τώρα. Ας πούμε, είχαμε στην Ιρλανδία ε, με την τράπεζα αυτή που κατέρευσε και τα προβλήματα που δημιούργησε στον Ιρλανδικό προϋπολογισμό, τότε δεν είχαμε καμία συμφωνία για κανένα PSI, για καμία συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και η συζήτηση μας πήρε 1,5 χρόνο πριν ε, ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Επομένως, είχαμε αυτές τις ad hoc αποφάσεις ε, είναι πολύ καλύτερο να ξέρουμε τι θα γίνεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Ούτως ώστε το μέλλον, όταν μια χώρα ζητάει ένα δάνειο ESM του από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας να κάνει μια ανάλυση ε, βιωσιμότητας το ESM και αν υπάρχει πρόβλημα ρευστότητα δεν θα γίνει αναδιάρθρωση. Το, η αναδιάρθρωση σημαίνει μαζική ε, παρέμβαση στα δικαιώματα ας πούμε, των ιδιωτών. Και όταν έχει πρόβλημα απλώ ρευστότητα, δεν υπάρχει λόγο να παρέμβει. Αν υπάρχει όμω θέμα φερεγκιότητα, είναι απαραίτητη η αναδιάρθρωση. Επομένω, πρέπει να γίνει πρώτα μια σοβαρή ανάλυση για να περάσουμε στην αναδιάρθρωση. Επίση, οι ρήτρε συλλογική δράση θα πρέπει να ενισχυθούν. Ενισχύθηκαν μια φορά το 2012. Έγιναν καλέ προτάσει ε, για να πάμε ακόμα πιο πέρα για είναι πολύ πιο δύσκολο να μπλοκάρουν κάποιοι την αναδιάρθρωση και το ESM θα μπορούσε να παίξει το ρόλο του διαμεσολαβητή για να φέρει γύρω από το τραπέζι τους συμμετέχοντες για να βρεθεί μια δίκαιη λύση για όλους. Ε, Αυτό όταν μιλάω για ένα πλαίσιο αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους. Ε, επιλέγω τη λέξη πλαίσιο πολύ προσεκτικά, όχι μηχανισμό, όχι αυτό που συζητούσαμε στο Δούνου του πριν από 15 χρόνια, που θα ήταν πιο άκαμπτο με αυτόματους κανόνες. Το πλαίσιο είναι, ξεκαθαρίζει τα πράγματα, είναι πιο προβλέψιμη κατάσταση και θα ήταν χρήσιμη, χρήσιμο συμπλήρωμα σε αυτά που συζητάμε σήμερα που είναι η δημοσιονομική ικανότητα. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε εσείς. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις. Για έξι σημεία Πρώτον, η σχέση μεταξύ ενωσιακού προπολογισμού και προπολογισμού ευρωζώνης. Νομίζω ότι υπάρχει μια κοινή ανησυχία που είναι η άκουση των κινδύνων. Ζούμε σε έναν κόσμο πιο αβέβαιο και κατ' αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα ποσοστό στον προπολογισμό που να προβλέπει αντιμετώπιση έκτακτων απρόβλεπτων περιστάσεων. Το ίδιο ισχύει και για τον ε, ενδεχόμενο προεπλισμό της Ευρωζώνης. Δεν θα μπω τώρα στη συζήτηση <clears throat> για το ποιο θα είναι το μέγεθος αυτού του προεπλογισμού. Αλλά αν είναι μικρός, ο προεπλογισμό θα πρέπει να εστιάσει τις πιο μεγάλες σοκ, που σημαίνει ότι στις περισσότερε περιπτώσει δεν θα χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια οικονομολόγοι γι' αυτό τείνουν να προτιμούν κάτι σχεδόν αυτόματο. Εσείς είπατε νομίζω. Ότι αν δεν έχουμε φορολογία δεν έχουμε αντιπροσώπευση και το ανάποδο. Άρα δεν έχουμε και ε, δαπάνες. Εγώ αυτό το αντιλαμβάνομαι. Γι' αυτό και λέω ότι προτιμούν πιο αυτόματο. Σε ό,τι αφορά το μέγεθος, Κάναμε κάποιες προσωμιώσεις με ένα μικρό προπολογισμό, εστιάζοντας σε μεγάλα σοκ, παραδείγματος χάρη ποσοστά ανεργίας που ανεβαίνουν πάνω από δύο ποσοστίες μονάδες. 0,25% του ΑΕΠ ανά έξτρα ποσοστία μονάδα ανεργίας. Από μακροοικονομικής πλευράς είναι αρκετά ε, μεγάλο το ποσό. Κάναμε κάποιες προσωμιώσεις. ως σημείο κίνησης, για να, γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό φόρο. 0,1% είναι η εισφορά ακατέτος. Αν ξεκινήσουμε το 99 φτάνουμε σε 70 δις το 2007 και το 2012 10 δις. Άρα δεν θα είχε εξαντληθεί το αποθεματικό αυτό με στην κρίση. Κύριε Ρέγκλινγκ, δεν φορά ποια είναι. Εμείς δεν μιλάμε για δάνεια, αλλά για επιχορηγήσεις. Ο δανεισμός είναι δουλειά του ESM, μακροχρόνια, ίσως και μακροπρόθεσμα στο μέλλον δάνεια. Εδώ εμείς μιλάμε για επιχορηγήσεις, που δεν αποπληρώνονται. Αλλιώς δεν έχει και νόημα. Γιατί περισσότερε χώρε δεν είναι αποκομμένε από τι αγορέ, μπορούν να δανειστούν. Άρα γιατί να υπάρχει αυτό το σχήμα. Πρέπει να είναι μια μεταφορά πίστος, όχι μόνη. Μόνο τη χρονιά που σημειώνει μεγάλη άνοδο η ανεργία. Μετά δεν προσφέρεται αυτό το πόσο δεν υπάρχει εξάντε λοιπόν εκ των προτέρων ε, μόνο εκ των υστέρων, γιατί δεν μπορεί να ξέρει κανεί πού θα χτυπήσει η ανεργία. Για τι χώρε που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη. Ακούστε, οι μακροοικονομικέ ανισορροπίες σε μια χώρα μπορεί να είναι συστημικές μόνο εντό Ευρωζώνης. Η μακροοικονομική κρίση σε μια χώρα μπορεί να πυροδοτήσει χρηματοοικονομική κρίση που να βάλει σε κίνδυνο την ίδια την Ευρωζώνη μόνο στην Ευρωζώνη. Όμω, αν είναι αυτή η χώρα, αν έχει κρίση μια χώρα εκτό Ευρωζώνη, επηρεάζει σίγουρα αρνητικά και την Ευρωζώνη, αλλά όχι μέσω νομισματικών διάβλων. Και εδώ μιλάμε για την ε, μη βιωσιμότητα του χρέους και μιλάμε για τα ποστά του ΑΕΠΑ. Uh, Σε ό,τι αφορά τι προκυκλικέ πολιτικέ, ναι, το 2009 συμφωνώ. Οι ευρωπαϊκέ δημοσιονομικέ ήταν αντικυκλικέ. Μετά όμω, το 2009-2012, ήταν προκυκλικέ που είχαμε το δεύτερο πρόβλημα. Και δεν είχαμε εργαλεία. Αν χρειαζόταν να ξαναερχίσουμε, αν είχαμε μια τρίτη βουτιά, πάλι δεν θα είχαμε ε, μέτρα να την αντιμετωπίσουμε. Πέμπτο σημείο. Συμφωνώ με την Περβάνς ότι το καλύτερο μέτρο είναι ένα επίδομα ανεργία. Επανασφάλιση, αν θέλετε, για μεγάλους κινδύνους. Αυτό είναι ουσιαστικά. Αυτό βοηθάει να έχουμε σταθεροποίηση. Δίνουμε δηλαδή σαν οικοκυριά που έχουν πρόβλημα ένα τσέκ, αν θέλετε, που μπορούν να το εξαργυρώσουν. Δεν υπάρχει καθυστέρηση. Πηγαίνει αμέσως το ποσό τον καταναλωτή. Γιατί με τι επενδύσει υπάρχει ο κίνδυνος. Με την καθυστέρηση να θέλει να είσαι αντικυκλικό, αλλά τελικά λόγω καθυστέρησης γίνεσαι προκυκλικό. Επίση τα χρήματα δοχετεύονται στο άτομο, το μεμονωμένο. Αν αυτό το άτομο αντιλαμβάνεται ότι τα χρήματα προέρχονται από την Ένωση, όπω το Έρασμο για παράδειγμα, πρέπει να προσπαθήσουμε να μιμηθούμε την επιτυχία του έρασμού. Γιατί βοηθάει να βελτιωθεί η ζωή του πολίτη. Απτά. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια επιφυλακτικότητα. Γι' αυτό σε ένα σύγγραμμα προτείνω μια ένωση απασχόληση, Jobs Union. Με κάποια μορφή σύγκλησης, επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, κινητικότητα, φορητότητα επιδομάτων, δικαιωμάτων και όχι μόνο συνταξιδοτικών δικαιωμάτων κτλ. κτλ. Μπορώ να σα δώσω λεπτομέρειες αργότερα. Και σύνδρομο Ντοβίλ τέλο. Για να το αποφύγουμε αυτό το σύνδρομο, σημαίνει ότι πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε αναταραχή στι αγορέ των κρατικών ομολόγων. Ποιο είναι το πρόβλημα. Αν ποτέ δεν λάβουμε υπόψη μα ότι θα μπορούσε να υπάρχει δυνατότητα αναδιάρθρωσης χρέου, θα προκύψει κάποια στιγμή πρόβλημα με τη συνθήκη. Εγώ δεν μπορώ αυτό να το δω ω μόνιμο, μόνιμη κατάσταση. Εμείς με την έκθεσή μας λέγαμε να μην εισαχθούν οι κανόνες. Τα junior bonds ας τα αφήσουμε έξω. Η βασική ιδέα είναι να μην έχουμε ενός κανόνες. Κάτι που θα έρχεται να προσθεθεί στα ήδη φυστάμενα μέτρα. Απλά να βρούμε τον τρόπο να εφαρμόσουμε αυτά που ισχύουν η ΕΚΤΑ όταν δεν έχει μια χώρα βιωσιμό χρέο, υποτίθεται δεν πρέπει να την ε, δανείζει. Το κάνει όμω. Το θέμα είναι πώ θα αλλάξουμε το σύστημα, ώστε να είναι δυνατόν οι υφιστάμενοι κανόνε να εφαρμόζονται. Αυτό. Σας εξήγησα τι γίνεται με τις εγγύσει, τα collateral, collaterals από τις τράπεζες. Έτσι μειώνουμε το κίνδυνο, δεν τον αυξάνουμε. Και χάρη στα άλλα στοιχεία επιμερισμού κινδύνου, πάλι μειώνεται ο κίνδυνος με τις αλλαγές αυτές. Και ο κίνδυνος για το δημόσιο χρέος και ο κίνδυνος για τη μετατροπή χρέους μειώνονται με τα νέα μέτρα αυτά. Ο κ. Φαμπρίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές για τις πολύ ε, ευφύς ερωτήσεις. Τρία σύντομα σχόλια. Το πρώτο, σε το σχεδιασμό και τη διακυβέρνηση της δημοσιονομικής ικανότητας που αφορά κυρίως αυτά που ο κύριο Μούρεσαν. Δεν μιλάω για το μέγεθος του προπολογισμού, οι οικονομολόγοι τα ξέρουν καλύτερα από μένα αυτά. Αλλά θα περιοριστώ στο κατά πόσον πρέπει να είναι μια γραμμή ε, στο πλαίσιο του ενωσιακού προβλησμού ή να είναι ένα ξεχωριστό προβλησμό. Από νομική πλευρά ε, είναι και τα δύο ε, εφικτά. Αντρετή κοστό. Υπάρχει το θέμα της ομοφωνίας, το είπα ο κ. Σαρτουή. Παρακαλώ, λίγο πιο αργά. Ναι, ναι, με συγχωρείτε. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα να έχουμε χωριστό προπολογισμό για την Ευρωζώνη, χωριστό δηλαδή από τον Ενωσιακό για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ομοφωνίας. Αλλά αντιλαμβάνομαι πόση μεγάλη σημασία έχει η ενότητα του ενωσιακού προπολογισμού. Και βέβαια αν έχουμε ξεχωριστή γραμμή στον προπολογισμό, τίθενται άλλα θέματα που έχουν να κάνουν τη διακυβέρνηση. Το είπα και στην παρουσίασή μου, νομίζω, ξεκάθαρα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει πλήρω στι αποφάσει που λαμβάνονται για τη δημοσιονομική ικανότητα. Αν είναι όμω ένα προπολογισμό για την Ευρωζώνη, θα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. West Lodge and Question λέγεται στον, στην νομοθεσία ότι μπορεί κράτη εκτό Ευρωζώνης να επηρεάζουν αυτά που συμβαίνουν εντός Ευρωζώνης. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει υποχρέωση για όλε τι χώρε να ενταχθούν στο ευρώ. Άρα το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει, έχει νόημα να συμμετέχει συνολικά στι διαδικασίε. Άλλο σημείο. Χρηματοδότηση του προπολογισμού. Από συνταγματική πλευρά είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα. Κύριο Μπέγκε και η κυρία Μάλετιτς αναφέρθηκαν στις ε, μεταφράσεις πιστώσεων από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Το θέμα είναι ότι όπω είναι σχεδιασμένο τώρα ο νησιακός περιορισμό βασίζεται ακριβώ στι εισφορέ των κρατών που αναδιανέμονται εν συνεχεία. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ψηφίσατε την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι δηλαδή παραβιάζει το σύστημα ιδιών πόρων ουσιαστικά τι διατάξει τη συνθήκη, το πνεύμα τη συνθήκη. Και το πνεύμα και το γράμμα παραβιάζει και δημιουργεί και ένα φαύλο κύκλο. <coughs> Γιατί Μπορεί κανείς να πει, οι ψηφοφόροι μου δίνουν χρήματα τα οποία πηγαίνουν αλλού, σε άλλες χώρες. Και αυτός παίρνει το σπόρο μεγάλων αντιπαραθέσεων μεταξύ των κρατών μελών. Ξέρουμε ότι ο ΕΣΕΜ βασίζεται στις εθνικές φορές. Και περίεργως τα κράτη-μέλη ε, επιβλέπουν την χορήγηση αυτών των κονδυλίων και θα ήταν περίεργο να πάμε σε μια κατεύθυνση να έχουμε αύξηση ιδιοπόρων, να μειώσουμε τον ΦΠΑ και το εθνικό στο εισόδημα και από το παραθυράκι όμως να τα ξαναφέρουμε μέσα χρησιμοποιώντας τα χρήματα του ESM και φτάνουμε έτσι ξανά στην αφετηρία, <clears throat> στην εκκίνηση. Πρέπει πάντως να αντιμετωπίσουμε ε, κατάμετα την πραγματικότητα για το θέμα της χρηματοδότησης αν όλοι ωφελούνται, θα πρέπει αυτή η πόρη να είναι το αποτέλεσμα του πλότου που δημιουργεί η Ένωση. Και όχι χρήματα τα οποία πηγαίνουν από τη... πληρώνει το ένα και τα παίρνει κάποιο άλλο. Για τον κύριο Χέις, που πράγματι εκπροσωπεί το Δουβλίνο. Συμφωνώ με τις ανησυχίες που εκφράστηκε Χέις για την έλλειψη όρεξης και βούλησης για αυτές τις αλλαγές. Από πλευράς είναι αναπόφευκτο αυτό η απόσταση του μένου Βασιλείου θα υποχρεώσει τα άλλα κράτη-μέλη να αναπροσαρμόσουν τι συνθήκε σε μια σειρά από διατάξει. Ήδη έχουμε μπει σε αυτή τη φάση, θα έλεγα. Γιατί η απόφαση περιδίων πόρων και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ουσιαστικά είναι περίπου το ίδιο με <clears throat> μια αλλαγή συνθήκη. Είναι δηλαδή σαν να έχουμε ήδη μπει στη διαδικασία τροποποίηση των συνθήκων. Και αυτό θα είναι ίσως μια ευκαιρία, ιδίως αν λάβουμε υπόψη το ψήφισμα που ψήφισατε πέρυσι για την αναθεώρηση της σύνδεξης Λισαβόνας που ίσως χρειαστεί για να έχουμε αυτό το πλαίσιο. Ευχαριστώ. Thank Κύριος Νιουνιέθ Φερέρ, θα περιοριστώ όσο μπορώ σε λίγες παρατηρήσεις. Η κυρία Γκρέσλα είπε κάτι σωστό αν μιλάμε για τα ίδια πράγματα. Νομίζω ότι ο ένα λέει το ένα, ο άλλο λέει το άλλο, ο τρίτο το παράλληλο. Μην ξεχνάτε ότι ο προπολογισμό σχεδιάζεται ω ένα επενδυτικό ε, προπολογισμό με επιπλέον ε, δυνατότητα σταθεροποίηση. Ε, από την επαγγελματική μου καριέρα ε, είδα ότι βλέπω να σχεδιάζουμε το ESM, το EFM το EMF μάλλον είναι ο ομιλητή, το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, ε, είναι φρικτό ω όνομα. Να μην αντιγράψουμε το δούνο του, Πάμε το πούμε κάπω αλλιώ. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να κάνουμε μια προσπάθεια σταθεροποίηση αλλού όμω. Αλλιώ αλλιώς τα βάζουμε όλα στον προπολογισμό και αυτό είναι επικίνδυνο. Γιατί θα υπάρχει αυτή η πίεση στον προπολογισμό και υπάρχει το πρόβλημα του μεγέθου του. Υπάρχει επίση μια ιδέα που συζητήθηκε και στο ΕΚΟΦΗΝ. Να έχουμε ένα τμήμα του προπολογισμού για τα κατεπήγοντα, για να αντιδρά, αντιδρούμε όταν υπάρχει κάποιο κατεπήγον. Ε, και απορρίφθηκε, γιατί τότε γίνεται πολύ μεγάλος ο προπολογισμός. Ε, γίνεται αυτή η συζήτηση λοιπόν. Πρέπει κάπου αλλού να βάλουμε λοιπόν τη σταθεροποίηση. Είναι δυνατόν αυτό το σύστημα ε, επιδομάτων ανεργία να μπει στο προπολογισμό. Ενδεχομένω, αλλά πρέπει να το ξαναδούμε. Για το μέγεθο του προπολογισμού τώρα. Νομίζω ότι ο ενωσιακό προπολογισμό, λόγω του περιορισμένου χαρακτήρα, θα πρέπει να περιοριστεί στο να χρηματοδοτήσει και να υποστηρίξει του εθνικού προπολογισμού που αγωνίζονται, που είναι πιο φτωχοί για να υλοποιήσουν πια του ε, ευρωπαϊκού στόχου. Και ζητώ, συγγνώμη που το φέρνω στο τραπέζι, αλλά έχουμε κάτι, έναν ελέφαντα εδώ πέρα που το βλέπουμε όλοι και δεν κανείς δεν μιλάει. Την κοινή αγροτική πολιτική. Ακόμα και αν τη μεταρρυθμίσετε. Ακόμα και αν δεν την αγγίξουμε. Αν αφήσουμε όλα ε, ίδια. Έχουμε τη νομική, τα νομικά ποσά, τις υποχρεώσεις κτλ. Αν την κρατήσουμε απαράλλαχτη. Πρέπει να δούμε πόσα λεφτά μετακινούνται. Είναι μόνο το 1 τέταρτο των χρημάτων της ΚΑΠ. Από όλα τα 45 δισεκατομμύρια, περίπου τα 30 δεν μετακινούνται καθόλου. Δεν υπάρχει μια μεταφορά όπω τα ταμεία συνοχή για να βοηθηθεί κάποιο. Έχουμε ε, μια κυκλική λειτουργία, α πούμε. Έτσι. Α πούμε, κοιτάξτε τη σχέση ας πούμε, του, της Γαλλίας με τις Βρυξέλλες ε, για τα γεωργικά, έτσι. Πάνε στην Γαλλία, γυρνά στις Βρυξέλλες, ας πούμε. Ε, κρατήστε κάποια λεφτά, α πούμε, στον προπολογισμό και τα υπόλοιπα απελευθερώστε τα για να κινούνται. Αν θέλετε να χρησιμοποιείτε πολιτικέ μέσα στον προπολογισμό, χρειάζεται χρηματοδότηση. Αλλιώ, εάν δεν αυξήσει τον προπολογισμό, μην χρηματοδοτείτε άλλε πολιτικέ. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν. Το θέμα είναι τι πρέπει να περνάει μέσω των Βρυξελών. Τελικά. Και δημόσια ε, οικονομική διαχείριση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε λογιστικά πρότυπα κτλ. Όλα αυτά είναι καλά για τι αναφορέ. Χρειαζόμαστε την ε, σταθερότητα. Αλλά προσοχή, προσοχή. Και υπάρχουν και χώρε που δεν το θέλουν. Γιατί μερικέ από αυτέ τι χώρε είναι πολύ πλούσιε. Φαίνονται θαυμάσιε, αλλά είναι εντελώ αδιαφανεί και τα λογιστικά του είναι εντελώ αδιαφανεί. Ε, η οίκη πιστοληπτική βαθμολόγηση ε, άρχισαν να κοιτάνε, ε, να βλέπουν τα λογιστικά. Ε, να βλέπουν τη σταθερότητα των γυναικών και αν αρχίσουμε των α, λογιστικών. Ε, μερικές... That maybe that movement... ε, μερικά λογιστικά μπορεί να μοιάζουν τέλεια σήμερα, αλλά μπορεί αύριο μεθαύριο να μην είναι, ας πούμε. Και το ξέρουν αυτό οι, οίκοι Πιστοποιητικής αξιολόγησης Δεν θέλω να ξαναντιμετωπίσουμε την, ελληνική κρίση α πούμε και να μας κατηγορήσουν πάλι ε, ότι δεν το προβλέψαμε. Ε, δεν προβλέψαμε την κατάρρευση χωρών που μοιάζαν ισχυρές. Ε, Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε μεταρρυθμίσει στις δημόσιες προμήθειες κτλ. Ε, για την δημόσια οικονομική διαχείριση. πολλά μπορούμε να κάνουμε με τις ε, αναφορές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αναφορέ αυτέ στη δημοσιονομική διαχείριση αλλά σε πολλές χώρες η δημοσιονομική διαχείριση δεν είναι σωστή και συχνά οι κανόνε του προπολογισμού δεν δίνουν κίνητρα, αλλά είναι αντικίνητρα για τις ε, αντικυκλικές πολιτικές τη χώρες, είναι αντικίνητρα για τις επενδύσεις τη χώρες και μιλάμε για καταστάσεις άλλη εποχή εποχής, του παρελθόντος. Και θα πρέπει αυτά τα, η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών να οδηγεί σε πραγματικό έλεγχο του χρήματο είναι φυσιο... Είναι φυσιολογικό. Θα πρέπει κάθε χώρα να εμπιστεύεται τις άλλε χώρε ότι δεν θα συμπεριφερθούν όπως να είναι και θα προκαλέσουν κρίση. Θέλουμε περισσότερη σοβαρή συμπεριφορά. Ναι, κατάρτιση, υποστήριξη των χωρών είναι σημαντικό, αλλά <laughs> Έχουμε στην κυριοστάτη ειδικού για τα λογιστικά, άλλους ειδικού για άλλα θέματα Κοιτάξτε πώς βοηθάμε την Πορτογαλία για να εισαγάγει τις ε, μεταρρυθμίσεις και την ε, διαχείριση των δημοσίων οικονομικών. Τα κοιτάω μεγάλο ενδιαφέρον. Ε, η δεύτερη χώρα που περνάει μέσα από αυτό είναι α, η Ελλάδα. Κατάλαβαν ότι πρέπει να αλλάξουν τα, την κατάστασή τους και ο, ο Πρωθυπουργό ε, ανήγγειλε μια πλήρη μεταρρύθμιση των δημοσίων οικονομικών φανταστικά νέα. Ίσως θα πρέπει να δούμε πώς το κάνουν. Και υπάρχει υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είναι τόσο ε, αδιαφανή η κατάσταση που κανένα δεν ξέρει πώ γίνεται, αλλά γίνεται. Και είναι τέλειο που γίνεται. Αυτά ευχαριστώ. Thank you very much. There were some questions also for the Commission. Για την Κομισιόν, ακούστε κάποιε ερωτήσει, θέλετε να απαντήσετε. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ. Ε, μας δίδεται η ευκαιρία και εμάς να απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις. Νομίζω η συζήτηση ήταν εξαιρετικά ε, χρήσιμη και ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι την Επιτροπή Προπολογισμών και Οικονομικών που διοργάνωσε αυτή τη ε, συζήτηση. Κανείς νομίζω δεν αμφισβητεί την ιδέα ότι η Ευρωζώνη χρειάζεται ε, μια λειτουργία δημοσιονομικής σταθεροποίησης. Ε, και αυτό καταδείχθηκε στη συζήτηση ότι είναι αναγκαιότητα για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ. Δεν άκουσα κανέναν να αμφισβητήσει αυτό το θέμα. Το θέμα είναι το πώς θα το πετύχουμε. Θα ήθελα δύο ερωτήσεις να ε, συζητήσω, τις οποίες απίφθηνε ο κύριος Γουαλτιέρη κατευθείαν. Πρώτον, ο ρόλος ε, του ESM μελλοντικού νομισματικού ταμείου για τη σταθεροποίηση και ο κύριος Ρέκλινγκ επίσης το ανέφερε. Εμείς ήδη εισηγηθήκαμε το Δεκέμβριο ότι ναι, το Μεντολοντικό Νομισματικό Ταμείο θα πρέπει να δημιουργήσει μια, ένα πιστοτικό όριο που θα πρέπει να ε, λειτουργεί ως ε, σταθεροποιητής. Και αυτό θα πρέπει να στηρίζεται ε, με εγγυήσεις μέσα από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Αυτό όμως έχει νόημα μόνο εάν οι δύο πυλώνες, ο Ευρωπαϊκός Προπολογισμός και το μελλοντικό IMF, είναι συνεκτικά και συνεπή σε ό,τι αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα κριτήρια ενεργοποίησης και επίσης υπάρχει και ένα θέμα διακυβέρνησης. Φτάνει ε, το ESM να παραμένει ένας διακυβερνητικός φορέας Εάν αυτή η θεραπεία, η λειτουργία θεραπείας δημιουργηθεί στα πλαίσια του τερέχοντος ESM, που είναι διακυβερνητικό σώμα, αυτό υπόκειται στην, στον κανόνα της ομοφωνίας. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το εξετάσουμε σε αυτό το πλαίσιο. Το δεύτερο σημείο που ε, ρωτήσατε ήταν το, το περιβόητο σύνδρομο Ντοβίλ, και όλη αυτή η συζήτηση για την αναδιάρθρωση δημοσίου χρέους. Θα πρέπει να είμαστε απόλυτα καθαροί σε αυτό και ξεκάθαροι. Δεν είμαστε υπέρ οτιδήποτε που θα γίνεται αυτόματα. Δεν είμαστε υπέρ κάποιες λειτουργίας που θα αποκλίνει από τις καλά εδρεωμένες πρακτικές του Δουνουτού που είναι περίπτωση κατά περίπτωση και ε, ε, βιωσιμότητας της κάθε χώρας. Δεν χρειαζόμαστε μηχανισμό να διόρθωση του δημόσιου χρέους και συμφωνούμε απόλυτα με τον Κλάους Ρέκλινγκ επ' αυτού. Το τελευταίο σημείο όμως είναι ότι μια συζήτηση στο θέμα αυτό ε, δύσκολο μπορεί να δει πώς μπορεί να το αποσυνδέσουμε από τον τομέα των τραπεζών. Θα πρέπει ε, μια τέτοια συζήτηση θα πρέπει να λάβει χώρα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ε, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης και ιδιαίτερα της ε, θέσπισης ε, της εγγύησης των καταθέσεων. Αν το κάνουμε ξεχωριστά θα μπορούσε να ήταν κάτι πολύ επικίνδυνο. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. Εισηγητές, κύριε Μπέκερ. Σύντομα κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ τους εμπειρογνώμονες που μίλησαν σήμερα ειδικά ε, τις συμβολές που μας δώσατε με κάποια πολύ ε, ενδιαφέροντα ε, στοιχεία που θα τα δούμε στις μελλοντικές ε, διαπραγματεύσεις. ο θέμα αρχής είναι καλό που αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία πάει προς αυτή την κατεύθυνση ότι χρειαζόμαστε μία δημοσιονομική ικανότητα με το μετασχηματισμό του ESF σε ένα είδους νομισματικό τομέα. Η... Δεν έχει συζητηθεί ακόμη η, κυβερνητική δια... δομή της διακυβέρνησης. Αφετέρου όμω, μετά από αυτές τις ακροάσεις και τα εργαστήρια, ε, και με αυτά που ανέφερε ο κύριο Νούνες είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε, να μην το ξεχάσουμε σε αυτό το πλαίσιο. Είναι σημαντικό να έχουμε κάποιες ε, δυνατότητες χρηματοδότησης αυτής της ε, δημοσιονομικής ικανότητας, ευρύτερε ε, δυνατότητες να καταλήξουμε σε συμφωνία με τα κράτη-μέλη και να μην επικεντρωνόμαστε μόνο σε ένα στοιχείο, αλλά να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα των συνθήκών μας που είναι διαθέσιμα σε εμά. ξανα... Δεν πρέπει να ξαναφεύρουμε τις συνθήκες και να περιμένουμε άλλα 9-10 χρόνια. Είναι, ήρθε η ώρα να δράσουμε και να δείξουμε ότι ως Κοινοβούλιο είμαστε διατεθειμένοι να σταθεροποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και να κάνουμε ό,τι καλύτερο ε, με προδραστικό τρόπο, να έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία, ε, γιατί μπορεί να προκύψουν κρίσεις όπως έχει συζητήσει. Ευχαριστώ. Πρέπει περάσει. Βλέπετε, από αυτά που σας είπαμε εκεί δύο, ότι το πνεύμα της έκθεσης είναι ζωντανό. Έτσι θα συνεχίσουμε, αν χρειαστεί. Θα σχολιασω για δύο-τρία πράγματα. Καταρχάς, για την αναδιάρθρωση του χρέους. Όλοι ε, συμφωνώ ότι μερικές φορές το χρέος γίνεται δυσβάσταχτο το επίπεδο του χρέους γίνεται δυσβάσταχτο. Μια απλή ιδέα θα ήταν να το διαγράψεις ή να το διαρθρώσεις. Αλλά αυτό έχει κόστος όχι μόνο για τη χώρα που πλήττεται από αυτό το μέτρο, αλλά και για την Ευρωζώνη συνολικά. Γιατί η χώρα η οποία θα πληγεί από την αναδιάρθρωση αυτή, θα επηρεαστεί, θα χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο για να ανακάμψει από ότι αν είχε ακολουθήσει άλλη ατραπό. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα. Είχαμε όλη αυτή τη συζήτηση για την αναδιάρθρωση του χρέους χωρίς να εξετάσουμε τι σημαίνει σε οικονομικούς όρου. Αλλά και για την Ευρωζώνη τι θα σημάνει. Δεύτερον, ο Ζωζέ Λεάνδρο της Κομισιόν είπε κάποια πράγματα. Χαίρομαι που μίλησε για το θέμα της αυτόματης διαδικασίας σταθεροποίησης. Από την έκθεση του Κοινοβουλίου έχουμε διδαχθεί κάποια πράγματα για αυτή τη λειτουργία σταθεροποίησης. Σε ό,τι αφορά το μέγεθος του προϋπολογισμού, να σας υπενθυμίσω κάποια νούμερα που δεν τα ξέρει το κοινό, δεν τα θυμάται το κοινό. Αλλά το μέγεθος του ESM, του Μηχανισμού Σταθερότητας, ε, η δανειοδοτική ικανότητα του ESM είναι 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Ε, το διαθέσιμο ρευτό είναι 772 δισεκατομμύρια. Ε, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης είναι 900 δισεκατομμύρια ευρώ. Σημαίνει ότι η δανειοδοτική ικανότητα του ESM είναι 5,05% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε. Ε, πέρα από τα θέματα των επενδύσεων, πέρα από τα θέματα του μηχανισμού σταθεροποίησης. Ζητώ συγγνώμη που το θέτω τελευταία στιγμή, αλλά σας δίνει μια γεύση για το ότι εάν υπάρχει θέληση να κινηθούμε σε αυτήν την κατεύθυνση, υπάρχει περιθώριο χειρισμού και από τη συνθήκη. Πέρα από τα νούμερα που σας είπα, υπάρχει ένα θέμα, γιατί αυτό το δυναμικό βασίζεται στην εγγύηση, τις εγγύησεις που υπάρχουν στα χέρια των κρατών μελών. Και δεν φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσουν ε, τα κράτη-μέλη να μεταφέρουν αυτέ τι εγγύσει ε, και να τι εντάξουν στον οσιακό προπολογισμό. Μπορεί να γίνει κάποια στιγμή στο μέλλον, αλλά δεν πρέπει να γίνει τώρα. Γι' αυτό λοιπόν με τον πρόεδρο Γκουαλτιέρη και με άλλου πιέσαμε την Κομισιόν να αλλάξει την πρότασή της ε, για το ESM και να βασιστεί στο 352, δηλαδή να βασιστεί στο κοινοτικό κεκτημένο με αναμφισβήτητο τρόπο, ούτως ώστε να παντρεύσουμε την κοινοτική μέθοδο με την εγγύηση του ESM πέρα από τον προπολογισμό της Ευρωζώνης. Της Ε, για τις χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη. Προς το παρόν όλοι είναι πολύ ευγενείς και κανένας δεν μιλάει για την επίπτωση που θα έχει αυτό στο μέλλον της Ευρωζώνης. Αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη που δεν είναι στην Ευρωζώνη μπορούν να μπουν στην Τραπεζική Ένωση εθελοντικά. Φανταστείτε ότι μετά το Brexit θα πρέπει να υπάρχει ένα μεγάλο κίνητρο ε, of όλα τα κράτη-μέλη για όλα τα κράτη-μέλη για να ενταχθούν εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Μην ξεχνάμε ότι αυτό ήταν ο, ο στόχος μας, να συμφιλιώσουμε την Ευρωζώνη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν σημαίνει θα λυθούν όλα τα θέματα του προπολογισμού, αλλά πρέπει να είμαστε συνεπείς. Και θα βελτιώσουμε και την ακριβώς τη συνεπειά μας. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για μια άκρος χρήσιμη ενδιαφέρουσα ανταλλαγή όσο στο αυτό αυτού του εργαστηρίου. Δεν θα κάνω εγώ καταληκτικές παρατηρήσεις, ε, το έκαναν οι συγητές. Ένα μόνο θα πω. Γιατί θεωρεί το Κοινοβούλιο σημαντική την ενσωμάτωση του ESM στο νέο κοινοτικό πλαίσιο. Επειδή είναι ο Κλάους Ρέγκλινγκ, εδώ τα λέω. Δεν ξεχνάμε ότι το ESM το χρηματοδοτούν οι εθνικοί προπολογισμοί. Είναι αυτή η δύναμη πυρό που είπατε. Είναι διαφορετική λογική από αυτήν του νοσιακού προπολογισμού. Δεν ζητάμε την ίδια δημοκρατική εποπτεία, τον ίδιο δημοκρατικό έλεγχο με την Κομισιόν ε, και του φορεί τη. Αντιλαμβανόμαστε πλήρω ότι αν ενσωματωθεί θα είναι κάτι σαν ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο και όχι κάτι διαφορετικό μάλλον σαν μια, θα είναι σαν την Τράπεζα Επενδύσεων, ε, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και όχι σαν κάτι άλλο. Το θέμα είναι να διαπραγματευτούμε όρους. Τι θα γίνει όμως που τα κάτι μέλη είναι μέτοχοι, που δεν θα δεχτούν. Θεωρούμε ότι από θεσμικής πλευράς είναι σημαντικό να μπει στο νομικό πλαίσιο της Ένωσης ο ESM και νομίζω ότι αυτό μπορεί να συμφιλειωθεί με την πλήρη αυτονομία και ανεξαρτησία του ESM. Δεν είναι και κάτι διαφορετικό από τη σχή τώρα. Σε σας δεν μιλάω γιατί δεν είστε μέλος ε, απλά Πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι και στο γερμανικό συνασπισμό, στις δηλώσεις προγραμματικές μέσα. Είναι σημαντικό να το έχουν υπόψη. Would... Να μην χάσουμε αυτή τη δυνατότητα λοιπόν. Σημαντική επένδυση μακροπρόθεσμη και όχι μόνο βραχυπρόθεσμη για την Ευρώπη. Τώρα είναι η ώρα να το κάνουμε αυτό. Βέβαια τη συζήτηση θα τη συνεχίσουμε, αλλά χαίρομαι που βλέπω να υπάρχει ευρεία συνένεση ως προς το να μην έχουμε ένα μηχανισμό, ένα πλαίσιο που είναι σημαντικό και θα δούμε πώς θα λειτουργήσει βέβαια. Αυτά τα junior 5 ετών πάνω από δεν ξέρω εγώ τι, το βρήκα πολύ εγώ extravagant. Μα όταν μιλάμε για μία αναδιάρθρωση γίνεται αυτό. Αν χρειάζεται αναδιάρθρωση δεν μπορεί να μην υπάρχει. Δηλαδή, αν, δεν έχουμε, αν έχουμε μία βόμβα, μπορούμε να κάνουμε ότι δεν υπάρχει βόμβα. Όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν υπάρχει, υπάρχει βόμβα. Μην επιμένουμε λοιπόν γιατί δεν θα σημειώσουμε πρόοδο στο σύστημα διακυβέρνηση. E uh, uh, Και το σημαντικό ζήτημα δεν είναι ο Ζαν Αρτουή, αλλά πάντων για εσά στην Επιτροπή Προπολογισμού το θέμα είναι το μέγεθο του προπολογισμού. Εμεί ω ΕΚΟΝ σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην Επιτροπή για τους προπολογισμού γιατί θα γίνει τεράστια, θα δοθεί τεράστια μάχη. Ξέρουμε την άλλη τις δύο και ελπίζω ότι συζητήθηκε σήμερα να μας βοηθήσει να αποκρισταλώσουμε τις απόψεις μας και για τις προσεχείς συζητήσεις και να μην χάσουμε το παράθυρο αυτό ευκαιρίε για να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ.